Bueno, a ver, pido a los Λοιπόν, να ζητήσω από τους λίγους παριστάμενους να καθίσουν, διότι θα ξεκινήσουμε με την απογευματινή συνεδρίαση. Έχουμε καθυστερήσει ήδη από το πρωί, έχουμε μείνει πίσω στο πρόγραμμα. Καταρχάς έχουμε το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον προπολογισμό ε, για τον Αλία για το 2011. Ε, συντάκτρια είναι η κυρία Ρόντας, Ε, όπως γνωρίζετε, το λέω στην κυρία Ρόντους, ούτως ή άλλως ε, αυτή θα τα πει. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου των συναδέλφων από την πολιτική μου ομάδα γιατί βρίσκονται σε άλλη συνεδρίαση. Είμαι βέβαιη ότι κάποια στιγμή θα φανούν. Ζητώ συγγνώμη που βρίσκομαι εδώ μόνη μου να τα πω. Έχω ενημερώσει του συναδέλφου. Καταρχά κάποια πράγματα διαδικαστικά. Το Συμβούλιο επισήμω δεν έχει εγκρίνει την πρότασή του και πρέπει ακόμα να περάσει από την Κορεπέρ το θέμα. Από εκεί και πέρα, βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν 8 εβδομάδε χρόνο για να ετοιμάσουν τι ε, δικέ του γνωμοδοτήσει και εκεί φαντάζομαι ότι θα έχουμε και νέε ε, ε, τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε βάσει των στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το παρόν σχέδιο ε, έχει 14 τίτλους ε, για την αλληλεία, στις οποίους έχουμε περικοπές ε, και νομίζω ότι σε κάποιους τομείς θα πρέπει να δαπανούμε κάποια περισσότερα χρήματα. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τροπολογίες προκειμένου να προσπαθήσουμε να αποσύρουμε τις περικοπές που έχει προτείνει το Συμβούλιο. Τώρα, για τις πιο σημαντικές ε, περικοπές από πλευρά Συμβουλίου, για τις πιστώσει υποχρεώσεων. Το συμβόλαιο θέλει να περικόψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Λίας ε, ε, κατά 200.000 ευρώ, που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να προσλάβει νέο προσωπικό. Δεύτερον, ένα εκατομμύριο θα περικοπεί από την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον έλεγχο που ασκείται από τα κράτη-μέλη. Μια άλλη γραμμή προπολογισμού για το για την εποπτεία που ε, δίνεται στα κράτη-μέλη θα έχει μια σημαντική περικοπή, 70.000 ευρώ. Και επίσης έχουμε τεχνική βοήθεια, ε, διασκέψεις, διαρμηνία κλπ. Και εκεί θα έχουμε περικοπές, ε, περίπου 110.000 ευρώ και κάτι παραπάνω. Διοικητικό κόστος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την Επιτροπή συγγνώμη, ε, θα κοπούν κάποια στοιχεία και εδώ. Ε, εποπτεία της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας. Ε, νομίζω ότι ε, δεν θα πρέπει να γίνονται περικοπές εδώ, διότι τέτοιου είδους εποπτεία είναι αυτή που μας λείπει. Επίσης, θα πρέπει να αποπτεύονται οι δαπάνες στις επίσημες αλληλευτικές συμφωνίες και εκεί θα έχουμε περικοπές. Και προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει έξι άτομα τα οποία ασχολούνται με την υλοποίηση. Έγινε τεράστια, μια τεράστια περικοπή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Λίας, 39 εκατομμύρια ευρώ και η αιτιολογία ήταν ότι έγινε κακή χρήση των πόρων στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι το 2011 θα γίνεται καλύτερη διαχείριση των ε, πόρων και θα έχουμε καλύτερη ροή χρημάτων, αλλά θα προτείνουμε τροπολογίες επί του θέματος οι περικοπές του Συμβουλίου επί των σημείων αυτών δεν είναι αποδεκτέ από πλευρά μας. Ε, είμαι βέβαιη ότι συμφωνείτε κι εσείς. Και θα τα αναφέρω τα θέματα αυτά και στην Επιτροπή Προπολογισμών και καλό θα ήταν ίσω και κάποια άλλα μέλη της Επιτροπής μας να έρθουν σε επαφή με τους συναδέλφους από την πολιτική τους ομάδα που συμμετέχουν στην Επιτροπή Προπολογισμών και να τους ζητήσουν να πιέσουν και αυτοί επί του θέματος. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τους και οδησυχητές. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και φυσικά θα ψηφίσουμε το θέμα αυτό την πρώτη μέρα μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι για το χρονοδιάγραμμα, αλλά πραγματικά ε, περιμένω να έχουμε αγαστή συνεργασία. Αν ε, επικοινωνούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντατικά, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συντάκτρια γνωμοδότηση ε, αναφέρθηκε στι βασικέ προκλήσεις. Είμαι και εγώ μέλο τη Επιτροπή Προπολογισμού, επομένω, και εγώ ασχολούμαι με το ζήτημα αυτό. Θα μπορούσα να σα μιλήσω λοιπόν και εδώ, όπω το έχω κάνει και στην Επιτροπή Προπολογισμού σήμερα το πρωί ασχοληθήκαμε με τη θέση του Συμβουλίου. Δεν πρόκειται για την οριστική και επίσημη ακόμα θέση του Συμβουλίου. Είναι μόνο σε επίπεδο κορεπέρ. Αλλά μπορούμε από τώρα να δούμε πάνω κάτω πώς θα είναι η θέση τελική του Συμβουλίου. Σήμερα λοιπόν το πρωί έγινε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το πόσο σημαντικές τομές, περικοπές έχουν γίνει στον τομέα της ε, αλίας. Ήταν πολύ σημαντική λοιπόν ε, η συζήτηση και φαντάζομαι ότι θα έχουμε την υποστήριξη της Επιτροπής Προπολογισμού προκειμένου να καταφέρουμε να ανακτήσουμε σε πιο λογικά επίπεδα κάποιες από τις γραμμές του προπολογισμού για την αλία. Και θα είμαι προφανώ σε επαφή και με την κυρία Ρόντα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητε τροπολογίε και να καταφέρουμε να ανακτήσουμε τα απολεσθέντα αυτά ποσά. Βέβαια, διανύουμε μια οικονομική κρίση, ωστόσο η προσέγγιση του Συμβουλίου είναι αρκετά προβληματική και θα έλεγα σε γενικότερο επίπεδο ότι θα έχουμε πολύ δύσκολες συζητήσεις στο φθινόπωρο. Αυτό είχε γίνει και πέρυσι το φθινόπωρο, επί του προπολογισμού, στις επαφές που είχαμε με το Συμβούλιο. Αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Βλέπουμε ότι προβλέπονται περικοπές από το Συμβούλιο, όχι μόνο στον τομέα της αλίας, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Δεν είμαστε οι μόνοι, δηλαδή, που πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές περικοπές. Υπάρχουν και άλλοι τομείς με ανάλογες περικοπές σαν αυτές τις αλίες ή πολλές φορές και χειρότερες. Δεν προσβλέπω λοιπόν στι δύσκολε αυτέ διαπραγματεύσει του φθινοπόρου. Προσβλέπω στι καλοκαιρινέ διακοπέ που ελπίζω θα μα δώσουν απαραίτητη ενέργεια για να δώσουμε τη μάχη αυτή του φθινόπωρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριο Στίβενσον. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις αυτές. Η κυρία ρόντα κάνει μια εξαιρετική δουλειά και πραγματικά έχει υποβάλει πολύ καλές προτάσεις, οποίε μπορούμε να υποστηρίξουμε. Το δικό μου το κράτος προβλέπει και αυτό σημαντικές περικοπές όπως η Ισπανία και η Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς δεν είναι δημοφιλής πολιτική αυτή για οποιονδήποτε πολιτικό. Από την άλλη όμως, ο προπολογισμό μα για την κοινή αλευτική πολιτική αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα τη γενικότερη γεωργική πολιτική, όπου δίδεται μία μάχη για να υπερασπιστούμε και το τελευταίο ευρώ το οποίο απομένει στην πολιτική αυτή. Έχουμε πολλά ευρωπαϊκά ύδατα τα οποία υπεραλλιεύονται και στη συνέχεια μας λένε από το Συμβούλιο ότι θέλουν να μειώσουν τον προπολογισμό για τον έλεγχο και την εποπτεία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το μήνυμα το οποίο πρέπει να δώσουμε είναι ότι αν θέλετε πραγματικά έναν τομέα αλίας με ανθρώπους που μπορούν να εργαστούν σε αυτόν και αν θέλετε πραγματικέ ε, βιώσιμες περιφέρειες και παράκτιες περιοχές, δεν μπορείτε με αυτόν τον βάναυσο και επιθετικό τρόπο να μειώνετε τον προπολογισμό. Συμφωνώ λοιπόν με την προσέγγιση της κυρίας Ρόντας. Ναι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρόντουστ. Συμφωνώ απολύτως, διότι ουσιαστικά σε όλες τις γραμμές ε, του προπολογισμού είχαμε σημαντικές περικοπές. Με ανησυχούν ιδιαίτερα οι περικοπές ε, που σχετίζονται με τις πιστώσεις υποχρεώσεων ε, περισσότερο από τις ε, υποχρεώσεις πληρωμών, διότι πρώτα πρέπει να γίνεται η δέσμευση για να καταβληθούν οι πόροι. Και μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός, διότι έχουμε πάρα πολύ μικρό ε, προπολογισμό στην αλληλεία και είμαστε και στη φάση αναθεώρησης της κοινή ελευθερικής πολιτικής που σημαίνει ότι όλα αυτά τα θέματα διοικητικά, μεταρρυθμίσεις όπου έγιναν ε, περικοπές κατά 25 ή 50% είναι απαράδεκτες διότι πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει επιπλέον προσπάθεια με συνεδριάσεις για να συζητήσουμε τα θέματα της μεταρρύθμισης. Πέραν των διοικητικών δαπανών και των τεχνικών δαπανών που επισημάνθηκαν και που επιμένω ότι είναι πολύ ανησυχητικές, θα πρέπει να θεωρούμε διπλά σημαντικό το θέμα της εποπτείας, διότι εκεί έγιναν πολύ σημαντικές επιτροπές, κυρίως το 11.08.02 που αναφέρεται στους επιθεωρητές που έχουμε στις Βρυξέλλες, οι οποίοι μεταβαίνουν στα κράτη-μέλη για να κάνουν τους ελέγχους και εδώ ε, μειώθηκε κατά ένα πέμπτο προπολογισμό. Επίσης, μου φαίνεται πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Ρόντουστ για, την, ε, για τον οργανισμό εποπτείας, ε, διότι πράγματι ναι μεν περιορίστηκε κατά το ίδιο ποσοστό ο προπολογισμό όλων των ε, υπηρεσιών, αλλά τα καθήκοντα της υπηρεσίας ελέγχου είναι πολύ πιο σημαντικά και ο προπολογισμό είναι πολύ λιγότερος από αυτόν που έχουν οι υπηρεσίες. Έγινε λοιπόν πολύ σημαντική διάκριση και προκειμένου να δούμε το θέμα των ταμείων. όντω μειώθηκαν τα κονδύλια σε όλα τα ταμεία, αλλά το ποσοστό μείωση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας ήταν το πιο σημαντικό ποσοστό από όλα τα υπόλοιπα ταμεία. Ε, μου φαίνεται λοιπόν απαράδεκτο όταν το ταμείο ούτως ή άλλως ε, ψυχία δίνει σε σχέση με τα υπόλοιπα ταμεία. Και εδώ οι περικοπέ ήταν ιδιαίτερα έντονε. Συμφωνώ απολύτως λοιπόν με τις ε, θέσεις. Ε, δεν ξέρω αν είναι το σχέδιο προπολογισμού, άλλη συνθήκη της ισαβόνας αλλάζουμε και τις ορολογίες τώρα συνέχεια, αλλά αυτό το οποίο θεωρώ εγώ είναι ότι φέτο με τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχουμε χάσει εξουσία στα θέματα του προπολογισμού και στι μη υποχρεωτικέ δαπάνε, ε, στι οποίε ε, στο παρελθόν είχαμε τον τελευταίο λόγο ε, δεν έχουμε πλέον τον τελευταίο λόγο και είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε σε θέματα συνδιαλλαγέ για τα θέματα τη αλληλεγγύη και ελπίζω να μην χάσουμε όπω χάνουμε και σε πολλά άλλα σημεία. Ελπίζω εδώ να υπάρχει αλληλοϊποστήριξη και εγώ θα είμαι σε επιφυλακή για να μπορέσω να συνδράμω. Ο κύριος Φερέιρα. Να να ζητήσετε λόγο. Bon, de facto, parece que Σας ευχαριστώ. Δεν πρόκειται μόνο για την διοργανική συμφωνία. Δεν είναι μόνο η διοργανική συμφωνία τομέα στον οποίο χάνουμε τελικά. Από ό,τι φαίνεται χάνουμε αρκετά και στον προπολογισμό. Εδώ πέρα έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα. και νομίζω ότι πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε πολλέ δυσκολίε. Συμφωνώ με τι ανησυχίε που εξέφρασε η συντάκτρια τη γνωμοδότηση, ιδίω για το ζήτημα τη παρακολούθηση τη εποπτεία αλεία. Η εισηγήτρια αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε έναν προπολογισμό που ξεκινάει ούτω ή άλλω από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Πρόκειται για ένα δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη του πραγματικά τις ανάγκες του τομέα. Και αντί να δούμε κάποια βελτίωση, βλέπουμε επιδείνωση, βλέπουμε περαιτέρω περικοπές. Πέρα από τους αρχικούς περιορισμούς έχουμε και περαιτέρω περικοπές τώρα. Και δεν νομίζω ότι μας δίνεται πλέον μεγάλο περιθώριο ευελιξίας. Το πολιτές πρόγραμμα αναφορά δεν μα δίνει περιθώριο ευελιξία και βλέπουμε ότι μειώνεται και ο προπολογισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και δυστυχώ δεν το αναφέρετε στην έκθεση. Ενδεχομένω θα μπορούσε να το συμπεριλάβετε. Και αυτό έχει σχέση και με τα μέτρα παρέμβαση στην αγορά. Η ρύθμιση τη αγορά είναι πολύ σημαντική για τομεί που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι και για το μίσο που επηρεάζονται από μια σημαντική οικονομική και κοινωνική κρίση. Ακόμα και σε αλία μικρής κλίμακας, είναι τελικά τα μέτρα, τα παρεμβατικά της αγοράς που επιτρέπουν στην αλία αυτή να, να επιβιώσει. Το ότι έχουμε λοιπόν ήδη από μόνο του δεν αρκεί, ήδη στο παρελθόν είχαμε εντοπίσει πολλά εμπόδια και προβλήματα και διάφορα κενά, αν τώρα πρέπει επιπλέον να επομισθούμε και περικοπές του προπολογισμό, νομίζω ότι η κατάσταση γίνεται πραγματικά παράδεκτη. Παρόλα αυτά τα προβλήματα, τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκα, τα παρεμβατικά μέτρα δηλαδή για την αγορά, ήταν τα μόνα τα οποία επέτρεπαν στους μικρούς αλείς να μπορούν να συνεχίζουν να κάνουν και δουλειά τους. Τώρα, οι περικοπές και στα μέσα αυτά θα πρέπει να αποσυρθούν ή τουλάχιστον να τονίσουμε το ότι χρειαζόμαστε αυτά τα μέτρα αν μη τι άλλο, ας επιστρέψουμε στην κατάσταση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Eh, Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, Νομίζω ότι το επίπεδο συνενέσεως σε αυτή την Επιτροπή δείχνει ότι η κατάσταση είναι ε, σημαντική. Περιμέναμε ότι θα υπάρξουν περικοπές, αλλά το Συμβούλιο έκοψε 14 γραμμές του υπολογισμού, ε, εκ των οποίων 9 ε, επιχειρησιακές δεσμεύσεις και πληρωμές και ε, εκεί η κατάσταση είναι ε, ε, δραματική διότι μιλάμε για 240 εκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό στο, στην Επιτροπή Προπολογισμού του Συμβουλίου ελπίζαμε ότι θα μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι δεσμεύσεις για το 2010 και το 2011 προέβλεπε μία παρεμφερή κατάσταση με αυτή τη 2010. Οπότε ετοιμάσαμε με πλήρη ταχύτητα τον προϋπολογισμό του 2011 και ορισμένοι από την Επιτροπή έχουν ήδη τονίσει γιατί όλες αυτές οι περικοπές είναι τόσο σοβαρές διότι τα προγράμματα πρέπει να εφαρμόζονται σωστά. Πρέπει να παρακολουθούμε τα κράτη το Συμβούλιο προβλέπει μία μείωση 240.000 στην αντίστοιχη γραμμή, 240 ε, εκατομμυρίων στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού και ε, περικόπτει επίσης και τη συλλογή δεδομένων. Δηλαδή έτσι θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων στα κράτη-μέλη. Είναι μια ε, καλώς εννοούμενη δαπάνη, διότι διαφορετικά οι ε, δαπάνες θα μειωθούν στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα προτού δημιουργηθεί. Βεβαίως όσον αφορά το γραφείο στο Βίγο 310.000 ευρώ είναι ελάχιστα για ένα τέτοιο γραφείο το οποίο έχει συνολικά 58 υπαλλήλους, τέσσερις συμβασιούχους και ε, με τις περικοπές αυτές μειώνεται κατά τρία τέσσερα άτομα, το προσωπικό των 58 ατόμων που δεν είναι τόσο τεράστιο αλλά θα πρέπει να ε, τονίσουμε ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι με την χρήση των πόρων αυτών και το Συμβούλιο έχουν μία γραπτή διαδικασία η οποία εξελίσσεται δηλαδή η πρόταση θα υιοθετηθεί στο Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου δεν περιμένω αλλαγές των αριθμών που ανακοινώθηκαν σήμερα στη συνεδρίαση. Πιστεύω ότι οι αριθμοί αυτοί θα ψηφιστούν στις 12 Αυγούστου και η Πρόεδρος είπε ότι είναι η πρώτη ε, χρονιά που θα έχουμε τη διαδικασία προϋπολογισμού ο, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας με συνδιαλλαγή σε τρεις εβδομάδες και εκεί ε, θα υπάρξουν διάφορες ρυθμίσεις, διάφορα παζάρια οπότε θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τη βοήθεια ε, του Επιτροπής σας για να αποκαταστήσουμε τον αρχικό προϋπολογισμό. Ε, Yeah, then... Ωραία τότε θέλω να ευχαριστήσω και είμαι ενθουσιασμένη με την αντίδραση της Επιτροπής διότι μόνο από κοινού θα είμαστε ισχυροί και θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Να βασιστείτε ότι εγώ θα κάνω ό,τι μου είναι δυνατόν ώστε να εξαλειφθεί αυτή η περικοπή. Ήδη επί τις εβδομάδες και μήνες δουλεύω σκληρά διότι είχα αντιληφθεί ότι η οικονομική κρίση θα ε, έχει αντίκτυπο και ε, στον προπολογισμό. Έχω κάνει πολλές συζητήσεις με τους αρμοδίους και τους είπα ότι χρειαζόμαστε όλα αυτά τα χρήματα για να ενισχύσουμε τους ελέγχους και να μην τους αποδυναμώνουμε. Και ε, υπάρχει 88% υπεραλία στις αλληλευτικές περιοχές μας, οπότε χρειαζόμαστε περισσότερες και όχι λιγότερους πόρους. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας παρακαλώ και εσείς τις πολιτικές σας ομάδες πρέπει να συζητήσετε με τους συναδέλφους διότι η Επιτροπή Προϋπολογισμού ήδη έχει τονίσει ότι υπάρχει κάποια ευαισθησία επί του θέματος και ελπίζω να τα καταφέρουμε στο τέλος. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρόντουστ. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών για τον προπολογισμό και για το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Ρόντους 20 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, ψηφοφορία στην Επιτροπή 30 Αυγούστου και ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών 28 με 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος. Θεωρώ λοιπόν λήξαν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 14 μία έκθεση για θέματα χρηματοδότησης και πάλι. Η συγκητή είναι ο κύριος Φερέιρα και έχουμε μία τροποποίηση του κανονισμού 861 του 2006, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται όλα όσα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Ο κύριος Φερέιρα είναι ο εισηγητής και θα μας εξηγήσει αυτή την ε, απλούστευση του κανονισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει και τη σύμφωνη γνώμη. Α, η αρχική παρουσίαση, συγγνώμη, θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ακούσουμε λοιπόν την αρχική πρόταση και πάλι ο κύριος ε, Τζόνσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως εξηγήσατε, αυτή είναι μία πρόταση να αλλάξουμε τον κανονισμό του Συμβουλίου 861 του 2006 που αναφέρεται ε, σε ένα δημοσιονομικό στοιχείο και μέσο το οποίο αποτελεί ένα από τα δύο βασικά μέσα χρηματοδοτήσεως της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Με το δεύτερο λοιπόν αυτό στοιχείο συγκεντρώνουμε τέσσερις ε, ενέργειες που καλύπτουν μεταξύ άλλων την διακυβέρνηση, τις επιστημονικές συμβουλές και την εφαρμογή και παρακολούθηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Για να ολοκληρώσω την εικόνα των δημοσιονομικών μέσων που έχουμε, έχουμε και ένα μικρό κανονισμό, ο οποίος ε, καλύπτει την στήριξη στις απόμακρες περιοχές και μια κοινή οργάνωση αγοράς για τα αλληλευτικά προϊόντα. Θα έπρεπε να σας πω σχετικά με το δεύτερο αυτό μέσο ότι είναι μία από τις ε, ε, μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να χρωματοδοτήσουμε και συμπληρώνεται από άλλους κανονισμούς και αποφάσεις του Συμβουλίου. Η τροπολογία την οποία έχουμε είναι μία σύντομη ε, τροπολογία με περιορισμένη φιλοδοξία ουσιαστικά προσπαθούμε απλούστατα να βάλουμε κάποια τάξη στην κατάσταση και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το δεύτερο αυτό στοιχείο είναι συνεκτικό και συνάδει με την υπόλοιπη νομοθεσία που αναφέρεται στο ίδιο θέμα. Από όταν λοιπόν εφαρμόστηκε αυτό το δεύτερο μέσο, είδαμε ότι υπήρξαν και νέες μέθοδοι, ε, πράγμα το οποίο ε, δείχνει πώς ε, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και πώς πρέπει να οργανωθούν τα χρηματοδοτικά μέσα. Θα πρέπει κάπως να προσαρμόσουμε το δεύτερο αυτό εργαλείο για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες τις οποίες πρέπει να καλύψει. Και ορισμένες αλλαγές τις οποίες θέλουμε να εφαρμόσουμε είναι μέτρα που διευκρινίζουν όπου είναι αναγκαίο το ε, θέμα το οποίο θέλουμε να χρηματοδοτήσουν. Επίσης προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση ορισμένων άρθρων στο δεύτερο αυτό στοιχείο. Αυτό προτείνουμε λοιπόν δεν αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο μέσο αυτό, ούτε ε, αλλάζει τα μέσα τα οποία προσπαθούμε να ε, διατυπώσουμε δεν έχει επιπλέον καμία δημοσιονομική επίπτωση για τον προπολογισμό. Απλούστατα η τροπολογία αποβλέπει να ε, διαμορφώσουμε καλύτερα τα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται στο χρηματοδοτικό κανονισμό, ιδίω ε, σχετικά με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν το 2006, διότι το σύνολο του προπολογισμού του θέματο είναι 6 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2009 ε, ήταν ε, εξ αυτών 268 εκατομμύρια ευρώ και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 είναι 271 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που θέλω να τονίσω και πάλι είναι ότι παρόλο που πρόκειται για μία απλώς βελτίωση, η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη, διότι αλλάζουμε διάφορα άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού, οπότε ε, είναι πολύ πιο εύκολο να διαβάσει κανείς τα, τις τροπολογίες από ότι να διαβάσει διαβάσει το αρχικό έγγραφο το οποίο είχε μία ροή. Ε, το Συμβούλιο έχει συζητήσει το θέμα αυτό σε επανειλημμένος ή στην ομάδα της ε, ε, αρμόδιας επιτροπής και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τομείς που καλύπτονται από αυτόν τον κανονισμό πρέπει να συγχωνευτούν και θα δούμε πώς διαμορφώνονται και αν αναφέρονται στο νομοθετικό πλαίσιο ή απλώς σε ε, μια τακτοποίηση των θεμάτων. Θα σας πω που έχουμε τις ε, λιγότερες αλλαγές στην πρόταση, διότι στο θέμα της ε, διεθνής, Διεθνούς Συμφωνίας ε, για την αλληλεία θέλουμε να διευκρινίσουμε την εμβέλεια του μέτρου. Δηλαδή, όταν μιλάμε για συνεργασίες στις Διεθνείς Αλληλευτικές Συμφωνίες, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι απλώς διμερείς, αλλά μπορεί να είναι και περιφερειακές και πολυμερείς. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε στον τομέα αυτό όσον αφορά τις οργανώσεις αλληλείας και το είδος συνεργασίας που μπορούμε να έχουμε μαζί τους. Στο παρελθόν ο κανονισμός μιλούσε για συνεργασία στον επιστημονικό τομέα ενώ μπορεί να υπάρξει και συνεργασία πέραν της επιστημονικής και θα θέλουμε αυτή η διάταξη να είναι σαφής στο σωστό πλαίσιο πλαίσιο. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, το δεύτερο τομέα που καλύπτει αυτός ο κανονισμός υπάρχουν ορισμένες, ε, ορισμένα σχόλια σχετικά με τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και τα περιφερειακά συμβουλευτικά συμβούλια τα οποία είχαν καταρτιστεί με απόφαση του Συμβουλίου ή είχαν δυνατότητα να καταρτιστούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του 2005 αλλά δεν ήταν συμβούλια τα οποία επιζητούσαν ένα γενικό κοινοτικό ευρωπαϊκό ε, συμφέρον. Έπρεπε λοιπόν να αλλάξουμε τη διατύπωση αυτή και να διευκρινίσουμε ότι τα συμβούλια αυτά θα τα χρηματοδοτούμε μόνο ε, στην πρώτη πενταετία. Έκτοτε όμως ε, θεωρούνται τα συμβούλια αυτά σαν θέμα γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η αλλαγή αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην νομοθεσία. Επιπλέον υπάρχουν ορισμένες μικρές αλλαγές ή στο εύρος των μέτρων που θέλουμε να αναφέρουμε για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μία κατάσταση όπου οι εκπρόσωποι συμμετέχουν στα συμβούλια και αναφέρουν πόσο συμμετέχουν, αλλά πρέπει να, να, να καλύψουν στην ε, εργασία τους και σε άλλου είδους συμβούλια και να εξηγήσουμε γιατί καλύπτουμε τα έξοδα της συμμετοχής στα συμβούλια αυτά. Αυτά είχα να προτείνω σχετικά με τη διακυβέρνηση. Στον τρίτο τομέα θέλω να αναφερθώ στη συλλογή δεδομένων, όπου υπάρχουν πολλές αλλαγές και αναφέρονται στο νομοθετικό πλαίσιο. Μάλιστα τέσσερις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που είναι σχετικές και πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο δεύτερο αυτό κανονισμό. Οπότε το 2008 που ανανεώσαμε το πλαίσιο ε, συλλογής δεδομένων ε, θέλουμε στο νέο κανονισμό να αντικατοπτρίζεται ότι στο δημοσιονομικό αυτό κανονισμό δεν μιλάμε μόνο για συλλογή δεδομένων αλλά και διαχείριση και χρήση. Όταν λοιπόν στηρίζουμε αυτές τις δραστηριότητες δεν στηρίζουμε μόνο τη συλλογή δεδομένων αλλά και τη διαχείριση και την χρήση που μπορεί να γίνει των δεδομένων αυτών. Το νέο πλαίσιο που εισήχθη το 2008 λέγει ότι καλύπτονται ε, οι διάφορες μεταβλητές ε, που αναφέρονται στην αλληλεία και στην υδατοκαλλιέργεια και θέλουμε αυτή η πτυχή να καλύπτεται στον κανονισμό. Τέλος, ε, στο νέο πλαίσιο του 2008 λέγεται Σαφώ σαφώς ποια είναι τα προγράμματα που μπορούν να αναλάβουν τα κράτη-μέλη για τη συλλογή δεδομένων και αυτά είναι τα στοιχεία που μπορούμε να στηρίξουμε και πρέπει ορισμένοι ορισμοί να αναφερθούν επίσης στο πλαίσιο αυτό. Τέλος, η άλλη αλλαγή που απορρέει από την αλλαγή αυτή αναφέρεται στις διαδικασίες προγραμματισμού που έχουν αναθεωρηθεί το 2008 και πρέπει τώρα ε, να νομοθετηθεί ανάλογα. Υπάρχουν και ορισμένοι ορισμένες ε, τροποποιήσεις οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στην αλλαγή των αναγκών και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε στις διεθνείς οργανώσεις οι οποίες αξιολογούν τα αποθέματα, πράγματα που γίνεται μέσω του ISIS και συλλέγουμε στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για να διατυπώσουμε πολιτικές. Έχουμε όμως και κάποιο πρόβλημα. Πολλές φορές αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συμβληθούμε με την ΆΙΣΙΣ και να τους ζητήσουμε να κάνουν κάτι συγκεκριμένο για λογαριασμό μας. Η τωρινή διατύπωση της νομοθεσίας δεν μας επιτρέπει να υπογράψουμε ε, μία σύμβαση δημοσίων αγορών και θα πρέπει να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το κείμενο για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την πτυχή. Τέλος, το τελευταίο θέμα που έχουμε σχετικά με τη συλλογή δεδομένων αναφέρεται στη διευκρίνηση που είναι αναγκαία, διότι το προηγούμενο πλαίσιο αναφερόταν στο 2007 και είχε καταργηθεί όταν ανελήφθησαν τα νέα μέτρα, τα οποία όμως δεν καλύπτουν κάλυπταν τις συγκεκριμένες πτυχές και έτσι τώρα ε, δεν έχουμε μεν προβλήματα με την απόφαση του 2008 για το 2009 και το 2010 έχουμε όμως προβλήματα για το 2007 και το 2008 ε, ίσως δεν είναι τόσο ουσιαστικό γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανόνες αλλά θέλουμε να υπάρχει νομική βεβαιότητα ότι οι, κατάλο... οι κανόνες τους οποίους εφαρμόζουμε ισχύουν και για το 2007 και για το 2008 και να μην υπάρχει ένα νομικό κανό. Τέλος, ε, αναφέρομαι στην εφαρμογή, όπου υπάρχουν ορισμένες αλλαγές σχετικά με τα μέτρα τα οποία πρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Αυτές οι τροποποιήσεις έχουν σχέση με την ε, ορθή οικονομική ε, διαχείριση. Προσπαθούμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη ή να τους καθορίσουμε μία ημερομηνία για να καταρτήσουν το πρόγραμμα πριν από κάποια ημερομηνία. Δηλαδή ε, είτε στις 31 του Ιανουαρίου ή μέχρι το τέλος του έτους που θα χρηματοδοτήσουμε ε, και θα πρέπει να προπορεύονται κατά τρεις μήνες για να μπορέσουν να περάσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να περάσουν από την Επιτροπολογία και ε, τελειώνει σχεδόν το έτος όταν μπορούμε να διατυπώσουμε τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες. Θέλαμε λοιπόν να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε καλύτερα τα προγράμματα αυτά. Και υπάρχουν και ορισμένε διατάξεις όπου προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις πληροφορίες που μα δίνουν τα κράτη όταν λαμβάνουν αυτά τα προγράμματα και εδώ αναφερόμαστε στα προγράμματα τα οποία εφαρμόζουν τα κράτη, αλλά και σε ορισμένα τα οποία ε, διατυπώνουν σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη. του ζητάμε πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επαληθεύσουμε τη χρήση που κάνουν των ε, μέσων ε, ελέγχου χρηματοδοτήσεως αυτών των προγραμμάτων. Δηλαδή όταν κάποιος μας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα για να χρηματοδοτήσουμε την αγορά ενός πλοίου ή ενός ε, αεροπλάνου θέλουμε να ξέρουμε πώς θα μετρήσουν τη χρήση που θα κάνουν διότι διαφορετικά όταν πηγαίνουμε επί τόπου δεν είναι εύκολο να επαληθεύσουμε εάν οι πόροι χρηματοδοτούνται όπως είχε δεσμευτεί το κράτος μέλος. Όσον αφορά τον έλεγχο, έχουμε κάποιες νέες διατάξεις που διευκρινίζουν περισσότερο τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου. Προσπαθούμε εδώ πέρα να κάνουμε μια συγκεκριμένη αναφορά στις δράσεις που πρέπει να χρηματοδοτηθούν μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τον έλεγχο. Θέλουμε να μπορούμε να χρηματοδοτούμε μέσα ελέγχου των σκαφών, αυτόματα μέσα ελέγχου, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και τη δημιουργία μια ιστοσελίδα που θα έχει να κάνει με τον έλεγχο τη αλεία. Επίσης, μία ακόμα διευκρίνηση έχουμε επιφέρει σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού όσον αφορά το ζήτημα του ελέγχου. Δεν μιλάμε πλέον για δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία έχουν δημοσίες υπαλλήλου που συνεργάζονται όμω με συμβασίουχους. Θέλουμε να καλύπτουμε πλέον όλο το προσωπικό, είτε πρόκειται για συμβασίουχους, είτε πρόκειται για μόνιμους δημοσίους υπαλλήλου. Επίσης, έχουμε αντικαταστήσει το irresponsible και illegal fishing με το responsible, illegal και unreported fishing. Έχουμε προσθέσει τον όρο unreported που δεν καταγράφεται. Προσπαθούμε λοιπόν να διευκρινίσουμε κάπως περισσότερο τα πράγματα, θέλουμε να τακτοποιήσουμε περισσότερο τα πράγματα. Δεν προσπαθούμε αυτή τη στιγμή μέσω των τροποποιήσεων αυτών να προεξοφλήσουμε το μέλλον της, τις μελλοντικέ αλλαγές που θα γίνουν στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Θέλουμε να καταφέρουμε γρήγορα να εγκρίνουμε τα νέα αυτά μέσα ή δυνατόν και σε πρώτη ανάγνωση, γιατί εφόσον πάρουμε γρήγορα με την έγκριση θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και τον, τον κανονισμό αυτό το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζόνσον, για τη της επεξήγησή σας. Ο κύριος Περέιρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εντελεχέστατη παρουσίασή της. Ο κανονισμός σαφώς είναι περίπλοκος και υπό το φως των τροπολογιών, αλλά η παρέμβαση της Επιτροπής ήταν πάρα πολύ σαφής και διευκρίνησε πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω και πάρα πολλά να προσθέσω αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα είπε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούν. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή αλλά και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για τα σχόλιά του διότι το κοινό μας μέλημα είναι να εξασφαλίσουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ ε, της ε, επιστήμης και των επαγγελματικών οργανώσεων δηλαδή των αλλιέων. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε τα ΡΑΞ, της ε, Περιφερειακές Επιτροπές και ε, στη συνέχεια ε, άρχισαν να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά όσον αφορά τις ε, αποφάσεις θα πρέπει να εμπλέκονται και οι επιτροπές αυτές για να μπορούμε να παρακολουθούμε την υγεία των, των αποθεμάτων αλληλείας και για να υπάρχουν υπάρχουν διαβουλεύσεις και γι' αυτό θα έπρεπε ε, σε κάθε συνεδρίαση ε, να μπορούν να εκπροσωπούνται τα συμβούλια αυτά, να καλύπτουμε τα έξοδά τους ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη αποδοχή και καλύτερη αποδοχή της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής αλληλείας να γνωρίζουν δηλαδή ποια είναι η κατάσταση όταν αλλιεύουμε τα αποθέματά μας και ποια είναι η κατάσταση διάσταση των θαλασσών μας και πιστεύω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να το επιτύχουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Ρόντας ε, και εγώ ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω μία σύντομη ερώτηση. Στο άρθρο 5 ε, ε, το οποίο τροποποιείται λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ζητά να διατυπώνονται οι δαπάνες των κρατών μελών με οικονομικά κριτήρια και αντελήφθη ότι θα υπάρξει συλλογή βιολογικών στοιχείων και δεδομένων. Θα θέλω όμως να ξέρω αν η Επιτροπή μπορεί να μας πει αν έχει καταρτήσει ένα κατάλογο προτεραιοτήτων σχετικά με τις ενέργειες αυτές. Ο κύριος yes, indeed, the commission. Πράγματι, η Επιτροπή επηρεάζει το θέμα αυτό. Η, τα προγράμματα συλλογή δεδομένων τεχνικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα κοινοτικά προγράμματα συλλογή δεδομένων και τα κοινοτικά προγράμματα καλύπτουν ε, ένα πολυετές ε, διάστημα και τα ε, εθνικά προγράμματα συλλογής δεδομένων ανταποκρίνονται στις απαιτήσει των κοινωτικών προγραμμάτων συλλογής δεδομένων. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Φερέιρα, θέλετε να δευτερολογήσετε. Όχι. Ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Και εδώ πρέπει να βάλουμε προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Όχι, όχι. Στις 29 Σεπτεμβρίου έχουμε παρουσίαση της έκθεσης. Ε, κλείνουμε λοιπόν με το σημείο 14 και τώρα περνάμε στο σημείο 17. Παρουσίασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ανακοίνωσής της σχετικά με τις ελευτικές δυνατότητες για το 2011. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πάτερσον. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Μια έξοχη καλοκαιρινή ημέρα και εμείς ετοιμάζουμε τις χειμερινές δραστηριότητες και κυρίως το Συμβούλιο. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τις επίσημες αλληλευτικές δυνατότητες για το 2011. Το έγγραφο είναι το COM 2241. Πρόκειται για ένα κείμενο για διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, ε, τα κράτη-μέλη και εσάς φυσικά για τα θέματα αυτά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για να προχωρήσει τα θέματα αυτά με διαφάνεια, για να δούμε τι γίνεται με τις αλληλευτικές δυνατότητες. Εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος ισότιμα για όλα τα κράτη-μέλη. Το πρώτο τμήμα αυτής της ανακοίνωσης έχει ε, μια αναδρομική ισχύ, εξετάζει από πού ξεκινάμε και προς τα πού οδεύουμε. Ε, θα σας ε, δώσω συνοπτικά κάποιες από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο έγγραφο. Καταρχάς, να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο αριθμός των αποθεμάτων που είναι γνωστά ότι δεν υπεραλλιεύονται ε, αυξάνεται. Το 2005 είχαμε δύο μόνο είδη, ενώ οι τελευταίες εκτιμήσεις είναι ότι έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Έχουμε λοιπόν μία μικρή αύξηση σε ένα μικρό ποσοστό αποθεμάτων, αλλά έχουμε δει βελτιώσει σε κάποια από τα αποθέματα τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης, εξετάζουμε πόσα ε, αποθέματα ή την χάνουν επιστημονική ε, γνωμοδότηση για να κλείσει η αλλιευσή τους. Ε, από το 2007 και μετά έχουμε μία μικρή μείωση ε, στις, οπι... Ε, γνωμοδοτήσεις οι οποίες προτείνουν να μην γίνεται καμία αλίευση. Αυτό αποδεικνύει βέβαια ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα τα οποία θα πρέπει να γίνουν και ακόμα έχουμε ένα 70% των αποθεμάτων που είναι εκτός των ασφαλών ορίων παρά το γεγονός ότι είχαμε μία μικρή μείωση τα τελευταία χρόνια, επομένως η μεγάλη πρόκληση παραμένει. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρθηκε ήδη είναι το γεγονό ότι η βάση πληροφοριών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, για την κοινή ελευθερική πολιτική, συγγνώμη, δεν βελτιώνεται. από το 2003 και μετά τα ποσοστά των στοιχείων που συλλέγονται είναι από 40 έως 50%. Σε γενικές γραμμές συλλέγουμε περισσότερα στοιχεία στη Μεσόγειο και ετοιμάζουμε περισσότερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ε, για την περιοχή. Υπάρχουν κάποιες βάσεις τις οποίες ε, θέλει να τηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, ε, η βιωσιμότητα από περιβαλλοντικής πλευράς που αναφέρεται στο βασικό κανονισμό για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις ποσοστώσεις σταθαρές στο μέτρο του δυνατού και να είναι συμβατές με τις περιβαλλοντικές απαιτήσει. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τα πολιετή σχέδια τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις διεθνείς δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει με τρίτες χώρες και φυσικά θα πρέπει να μειώσει ε, να μειωθεί η υπεραλίευση και να αποκατασταθούν κάποια είδη. Ε, όλα αυτά βασίζονται στη διεθνή συνένεση και στις επιστημονικές οδοτήσεις, δηλαδή του ISIS και του STCF. Ε, όπου βέβαια είναι πιο αβέβαια τα στοιχεία, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Το καινοτόμο στοιχείο φέτος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να κάνει ταχύτερες κινήσεις ε, για να εφαρμόσει το Wine. Υπάρχει η διάσκεψη ε, του Johannesburg του 2002 στην οποία συμφωνήθηκε ε, να ανασυσταθούν τα είδη ε, στο μέγιστο επιτρεπόμενο απόθεμα μέχρι το 2015 και για να επιτευχθεί αυτό μέχρι το 2015 πρέπει να αναλάβουμε δράση ήδη από τώρα, από το 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ζήτησε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να ανασταθούν τα αποθέματα μέχρι το 2015 και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε διαβούλευση με τα κράτη-μέλη ε, και τους ενδιαφερομένους επί του θέματος η μέθοδος εργασίας για τις αλληλευτικές δυνατότητες και τον σχετικό κανονισμό ως συνήθω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει μακροπρόθεσμα σχέδια βασισμένα στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και ζητά από τις Διεθνείς Επιτροπές να τους δίνουν στοιχεία για την κατάσταση των αποθεμάτων με βάση συγκεκριμένα σημεία και από εκεί και πέρα γίνεται ένας καταμερισμός των ε, ειδών σε 11 κατηγορίες. Παραδείγματο χάρη ε, από θέματα που ε, βασίζονται ε, στην αλλιεύση του συμβατά με το MSY και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα τα TAC εφαρμόζονται για όλα τα αποθέματα στις κατηγορίες αυτές. Δεν θα διατρέξω τις 11 κατηγορίες. Θα σας επισημάνω μόνο δύο αλλαγές οι οποίες ε, πρόκειται να γίνουν. Το πρώτο αφορά την ε, υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων σε σχέση με το MSY, με, το μέγιστο βιώσιμο με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και για να έχουμε έναν ε, ποσοστό θεμισιμότητας που να είναι συμβατό με αυτό που θέλουμε να έχουμε το 2015, αλλά να μην έχουμε μείωση περισσότερο του 25%. Επίσης υπάρχει ένας αντίστοιχος κανόνας ε, που δίνει ένα 30% ε, και δεν θα πρέπει να αλλάξει κάτι ε, κατά παραπάνω από 30%. Πρόκειται για αποθέματα τα οποία βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου. Υπάρχουν κάποια είδη για τα οποία δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τις συνέπειες των ε, αποθεμάτων και εκεί διατηρούμε τους ίδιους κανόνες αλλά εξακολουθούμε να ζητούμε τις νομοδοτήσεις του ISIS και του ISIS-TCF για μια προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να δούμε τι θα κάνουμε. Αν υπάρχει χαμηλότερη αλίευση ε, σε σχέση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μπορούμε να έχουμε αύξηση κατά 15%. Αν υπάρχει υπεραλίευση θα έχουμε μείωση κατά το αντίστοιχο ποσοστό. Εάν δεν υπάρχει καμία γνωμοδότηση για το κατά πόσον είναι συμβατό το είδος ε, με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τότε θα ισχύει μια αύξηση κατά 20% και ε, θα έχουμε και αντίστοιχα μείωση κατά 15% εάν θεωρούμε ότι υπάρχει διαφορά. Ε, και δεν αλλάζει τίποτα φυσικά εάν δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην αυθονία του είδους. Ε, αυτό γίνεται για είδη για τα οποία έχουμε λίγες βιολογικές πληροφορίες για το πώς έχουν οι τάσεις αλίευσης. Επίσης λάβαμε κάποιες νέες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από τον ICS τον Ιούνιο. Θα λάβουμε σύντομα και κάποιες γνωμοδοτήσεις από την ISTCF και θα προτείνουμε θα προετοιμάσουμε συγγνώμη, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα τάκια της ποσοστώσης τον Οκτώβριο. Αυτά όσον αφορά στην παρουσίασή μου για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Θα ήθελα τώρα να σταθώ σε τρία σημεία τα οποία συζητήθηκαν από τις περιφερειακές οργανώσεις Ελίας και ίσως έχουν κάποια σημασία εδώ. Αναφέρθηκαν κάποιες ανησυχίες για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ε, για το κατά πόσον είναι σε επιστημονικέ δρομοδοτήσει. Υπάρχει μια εκτίμηση και πόσο βασίζεται σε επιστημονικές γνωμοδοτησει Υπάρχει μια ανησυχία σε καποιου τομει για το κατά πόσον είναι ε, συγκεκριμένα αυτά τα στοιχεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις του FMSY που δίνονται από τους επιστήμονες είναι μία ένδειξη ως προς την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και από εκεί και πέρα προσαρμόζουμε τα TAC με βάση τις γνωμοδοτήσεις και τα αλλάζουμε σταδιακά όσο λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει επίσης ανησυχία για τη μεικτή αλία, στην οποία λιεύονται διάφορα είδη. Υπάρχουν κάποια τα οποία έχουν διαφορετικές παραμέτρους ε, ε, για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και εδώ θα θέλαμε να αναπτυχθούν κάποια τεχνικά μέτρα προκειμένου να επιτύχουμε ε, στοχευμένες αλίες για κάθε είδος. Ε, τέλος, κάποιες σκέψεις επί του θέματος Ορισμένε φορέ μπορούμε να έχουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση που να ισχύει για διαφορετικά είδη ανάλογα με τα στοιχεία που έχουμε για τα αποθέματα. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ μια προσαρμοσμένη μεθόδου που θα βασίζεται στι τρέχουσε εκτιμήσει και όπω αλλάζουν τα συστήματα, όπω αναπτύσσονται τα διάφορα περιβάλλοντα και θα αναθεωρούνται και οι ε, αποφάσεις μας. Αυτά ω προ την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πάτεσον για την περιγραφή της κατάστασης. Θα ήθελα να κάνω όμως και κάποιες παρατηρήσεις. Εμείς λάβαμε την ανακοίνωση αυτή μόνο στα ισπανικά. Αυτό ισχύει φαντάζομαι για κάθε μέλος επιτροπής Επιτροπή και θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο, γιατί δεν μπορούμε εμείς να προετοιμαστούμε, δεν μπορούμε να υποβάλουμε ερωτήσει. Υπάρχει κάποιο που το έλαβε σε κάποια άλλη γλώσσα ρώτησα κάποιου συναδέλφου και μου είπαν ότι μόνο σε Ισπανικά το λάβανε, εκτό μικροφώνου η παρέμβαση Προέδρου. Ε, Εδώ ο γραμματέα το έχει στα γαλλικά. Εδώ ήδη λοιπόν υπάρχει στα γαλλικά, φαντάζομαι ότι υπάρχουν σε όλε τι γλώσσε. Δεν ξέρω αν εσείς είχατε πρόβλημα στην πρόσβαση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει σε όλε τι γλώσσε. Δεν υφίσταται το κείμενο σε όλες τις γλώσσες. Ούτως ή άλλως μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ το κείμενο και να το πάρετε στη γλώσσα που θέλετε. Τόσο απλό είναι. Ε, τέλος πάντων, κύριε Λεβίνα, έχετε το λόγο.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 και εγώ είχα μόνο το ισπανικό κείμενο και δεν το διάβασα γιατί δεν ε, καταλαβαίνω καλά ισπανικά, αλλά ε, φίλοι μου μου ε, επισήμαναν δύο θέματα που θέλω να θέσω στην Επιτροπή. Καταρχήν επενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι προβλέπουν ότι μέχρι το 2015 θα υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο να συνάδει με την ε, σύγχρονη τεχνολογία. Ε, επίσης αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθούν να προωθήσουν ε, τα θέματα και ελπίζουν ότι το αποτέλεσμα εφέτος θα είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Και αντιλαμβάνομαι άλλωστε ότι για πολλά από θέματα ψαριών ε, δεν ε, υπάρχουν ε, επαρκή πόροι και πέραν αυτού έχω θέματα τα οποία με ενοχλούν παρόλο που συμφωνώ με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχει μια καλύτερη ε, τράπεζα δεδομένων. Αν είχαμε πιο αξιόπιστα στοιχεία, τότε η αποδοχή θα ήταν ίσως πολύ μεγαλύτερη. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχάς να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ανακοίνωσή της έχει ένα σημείο 4-2 που αναφέρεται στην αλληλευτική προσπάθεια και πάλι εδώ υποχρεούμε να σας πω ότι το θέμα της αλληλευτικής προσπάθειας δεν θεωρούμε ότι εμπίπτει στο άρθρο 43.3 και επομένως τα τάκες της ποσοσπώσης, οι αλευτικές ε, δυνατότητες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Πρόκειται για κάτι το οποίο επαναλάβαμε και πέρσι όταν καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τάκτη ποσοστώσεις βάσει της αλευτικής προσπάθειας ε, και θεωρούμε ότι δεν είναι τη αρμοδιότητα των τάκια των ποσοστώσεων. Δεν εμπίπτει στο άρθρο 43.3 και δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται λοιπόν εδώ η αλευτική προσπάθεια πέραν αυτού έχω και κάποιες άλλες ερωτήσεις και παρατηρήσεις να κάνω. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο στην τελευταία αξιολόγηση του ISIS ε, υπάρχουν κάποια αποθέματα τα οποία βασίζονται στο RMS ε, ή στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση όπως τη λέτε στα αγγλικά. Εκτός από κάποια συγκεκριμένα είδη, στα οποία στοχεύουμε συγκεκριμένα, όλα τα είδη στα οποία εστιάζει ο ISIS δεν έχουν ε, κάποια αξιολόγηση για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και ναι, μεν εξαιρετικά όλα αυτά τα οποία μα είπατε και οι στόχοι που θέτετε, αλλά αν δεν έχουμε μία αξιολόγηση τη νησιμότητας και τη μέγιστη βιώσιμης απόδοσης, τι παραμέτρου θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα, το FMAX ε, είναι κάτι αντίστοιχο με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αλλά δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι πότε θα έχουμε κάνει αξιολόγηση των αποθεμάτων βάσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Δεύτερον, κάτι το οποίο αναφέρατε κι εσεί πολυ... η αλία πολλαπλών ειδών. Ε, κάποιες ε, φορές ε, καθορίζεται μία μέγιστη βιώσιμη απόδοση βάσει κάποιου συγκεκριμένου αλλιεύμα, κάποιου είδους αλίας και όχι αναείδος. Ε, στα εναλία πολλαπλών ειδών θα ήταν πιο λογικό για να εξαλογίσουμε απορρίψεις και ούτω καθεξής. Και θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για την ερώτηση της κυρίας Ρόντους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω εγώ, βέβαια αυτές είναι ανεπίσημες πληροφορίες, στο Συμβούλιο Υπουργών λογικά έχει ξεκινήσει η συζήτηση και υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν δέχονται μείωση κάτω του 10% και υπάρχουν φυσικά μια σειρά από συμφέροντα που προασπίζεται ο καθένα και καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση είναι ακόμα ανοιχτή και τελικώ η απόφαση ως συνήθως θα είναι πολιτική. Κύριε Πάτερσον, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Αν ελπίζω ότι θα αλλάξουν φέτο τα πράγματα, είναι πάντα το ελπίζω αυτό. Και μάλιστα έχει δικαιολογηθεί η στάση μου αυτή στα τελευταία χρόνια. Αν δείτε για παράδειγμα στο έγγραφο, μπορείτε να δείτε μία σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα του Συμβουλίου και τα όσα μας παρουσιάζουν οι διεθνείς συμβουλευτικές επιτροπές. Βλέπετε εδώ πέρα ότι τα τάξα είναι πολύ ψηλότερα από αυτά τα οποία είχαν ε, προβλεφθεί στην αρχή. Βέβαια, έχουμε και μία μείωση και μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά την κατάρτιση των συνολικών επιτρομενών αλλιευμάτων για συγκεκριμένα Πιστεύω λοιπόν ότι η θετική αυτή τάση θα συνεχιστεί. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια βλέπει διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά τη συμπερίληψη της ελευτικής προσπάθειας εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και επικεντρωνόμαστε σε ελευτικές δυνατότητες και στην, στον τρόπο που συνδέονται με τις ποσοστώσεις. Ξέρουμε ότι ε, η ISIS έχει προσπαθήσει να καλύψει όπου είναι δυνατό όλα τα αποθέματα. Κάνει ότι καλύτερο δηλαδή μπορεί προκειμένου να υπολογίσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Επίσης για τα ε, είδη τα οποία μεταναστεύουν πολύ, δεν υπάρχουν όλα τα δεδομένα, ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα τον Οκτώβριο. Ζητάμε δεδομένα όσον αφορά τα πολλαπλά είδη, την πολλαπλή αλία, αν υπάρχουν δηλαδή κάποια κριτήρια τα οποία θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε συνολικά σε πάρα πολλά είδη και να υπολογίσουμε βάσει των κριτηρίων αυτών τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Επίσης, στην ε, Βόρεια Θάλασσα έχουμε ασχοληθεί με την γλώσσα συγκεκριμένα και πάλι βάσει δεδομένων που μας έχουν δοθεί από την ISIS και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια. Σας ευχαριστώ. Για την ελευθερική προσπάθεια μου απαντήσατε. πάντων δεν είναι για κανένα πρόβλημα, είναι γενικότερο πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα τα βάλω τώρα μαζί σα, ούτε θα σα υποχρεώσω να μα το εξηγήσετε εσεί αυτό το νομικό ζήτημα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πάτερσον. Θεωρούμε λοιπόν λήξα και αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης και συνεχίζουμε τώρα ε, με αυτά που είχαμε αφήσει σήμερα το πρωί το σημείο 12, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Χιλή για τη διατήρηση των αποθεμάτων ψηφία στο Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Κενό. Ο εισηγητή είναι ο κύριος Γκάλαγκερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, thank you, President, and thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ε, Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω τώρα για το ζήτημα αυτό. Η ίδια η πρόεδρος φαντάζομαι ότι γνωρίζει πολύ καλύτερα το θέμα από ότι εμείς. όλα αυτά, υποβάλλουμε κι εμείς μία γνωμοδότης για το ζήτημα αυτό. Φαντάζομαι πάντως ότι η δική σας εμπειρία που είχατε ως υπουργό σας επιτρέπει να έχετε πάρα πολλές γνώσεις για το ζήτημα αυτό. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τον Ισπανικό Σύλλογο και μας είχε ζητήσει να δούμε πώς μπορούν οι αλληλευτικοί στόλοι να έχουν πρόσβαση στα χωρικά ύδατα της Χιλής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να διευθετήσει το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η Χιλή στη συνέχεια έθεσε κάποια ερωτήματα που είχαν να κάνουν με την διευθέτηση διαφορών στα πλαίσια του δικαίου της θάλασσας σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών. Στις 19 ε, Δεκεμβρίου του 2000 ετέθη το ζήτημα της ε, εκμετάλλευσης ε, συγκεκριμένων ειδών στα χωρικά ύδατα της Χιλής και στη συνέχεια τον Ιανουάριο του 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Χιλή κατέληξαν σε μία προσωρινή συμφωνία όπου συμφώνησαν όλα τα συμβαλόμενα μέρη ότι θα υπάρχει μία παράλληλη αναστολή των ε, αποφάσεων που ε, είχαν ληφθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, καθώς επίσης και από το αρμόδιο δικαστήριο για τα θέματα της θάλασσας, για τα λευτικά θέματα. Τον Οκτώβριο συνέχεια του 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε μία απόφαση βάσει τη οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με τη Χιλή εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προκειμένου να φτάσουμε πλέον σε μια οριστική συμφωνία για το νέο πλαίσιο συνεργασία στον τομέα της αλίας και μετά από μερικού μήνε τον Οκτώβριο του 2008, καταφέρανε να καταλήξουν οι διαπραγματευτέ σε ένα τελικό κείμενο. Το Δεκέμβριο έπειτα του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο την έκβαση των διμερών τεχνικών συζητήσεων που γίνανε με τη Χιλή και οι οποίες λάβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2009 στη Νέα Υόρκη όπου βλέπουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τα ευρωπαϊκά σκάφη τα οποία επιθυμούν να λιεύσουν στα... στην περιοχή της Χιλής. Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2009, το ειδικό τμήμα του Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας αποφάσισε να ε, δώσει μια λύση στο ζήτημα αυτό μετά από αίτημα το οποίο είχε κάνει η Χιλή. Αποφάσισε να δούνε την πραγματική κατάσταση και τι γινόταν στην πράξη. Είχαν καταβληθεί άλλωστε πάρα πολλέ προσπάθειε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιληθεί το πρόβλημα. Δεν είχε επιληθεί για πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και στο τέλο τη δική μα θητεία, αλλά και στο τέλο τη επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, δεν, δεν θα έχουμε καταφέρει να βρούμε μια οριστική λύση στο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προσπάθησε να βρει μια λύση ήδη από το 2001 στα πλαίσια ενός μνημονίου το οποίο θα εφαρμοζόταν, εφαρμοζόταν προσωρινά. Η Χιλή δεν αντέδρασε όμως την προσπάθεια εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκείνη την εποχή και δεν υπήρχε κάποια βούληση συνεργασίας τελικά. Αυτή είναι μια σύντομη σφαιρική επισκόπηση των όσων συνέβησαν και των συστάσεων που έχω να κάνω προς την Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φράγκα για τη συμβολή της, καθώς επίσης και τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο εισηγητής, ο κύριος Σάντσες, η συμφωνία αυτή που από ό,τι βλέπω στις ε, υποσημειώσεις ξεκινάει από το 1999 όταν δημιουργήθηκε κάποια διαφορά για την πρόσβαση των ε, σκαφών που αλλιεύουν ξηφία και ε, υπευλήθη το ζήτημα στο σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Ε, στη συνέχεια με τη Χιλή προέκυψε μία διαφορά μεταξύ των, ε, όσων λέει ο ΠΟΕ και όσων λέει το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσης και από το 2000 και έκτοτε ε, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Υπάρχουν δύο θέματα βέβαια τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Καταρχάς το 2001 διακόπησαν όλες αυτές οι διαδικασίες και το δεύτερο είναι ότι από το 2003 υπάρχει μια συμφωνία διασύνδεσης με τη Χιλή και φυσικά έγινε κάποια ε, και υπάρχει ένα επίπεδο συνεννόησης για τα δύο θέματα τα οποία ήταν διαφιλονικούμενα. Το πρώτο αναφέρεται στην ε, διατήρηση των αποθεμάτων του Ξηφία και το δεύτερο είναι η πρόσβαση στους λιμένες της Χιλής. Ε, υπάρχει πρόσβαση σε τρία ε, λιμάνια, στο Περτορίκα, στο Αλταφαγώστα και ένα τρίτο και ε, αναφέρεται και το θέμα των αποθεμάτων του Ξηφία και ε, καθορίστηκε μια τεχνική επιτροπή για το άνοιγμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται διαβούλευση πολυμερός. Θεωρούμε λοιπόν ότι λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες και η προ... την πρόοδο που επετεύθηκε στο θέμα της επίλυσης της διαφοράς και το γεγονός ότι από πλευράς Χιλής απεσύρθη ε, η προσφυγή που είχε κάνει στο δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας, ε, θεωρώ ότι μπορούμε εμείς από πλευράς μας να ε, τηρήσουμε το άλλο τμήμα της συμφωνίας και έτσι να περατώσουμε μία διαφορά που αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν είναι πλέον δικαιολογημένη και πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για δύο συμβαλόμενα μέρη τα οποία έχουν υπογράψει μια συμφωνία σύνδεσης και δεν θα πρέπει να παρατείνουν άλλο αυτή τη διαφορά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να παρέμβω για να πω κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπε ο αγαπητός συνάδελφος. Πρώτον, η διαφορά με τη χιλή που ήδη αναλύθηκε έχει ως εξή. Τι είναι αυτό που παραβίασε και συνεχίζει να παραβιάζει η χιλή. Η χιλή παραβίασε την αρχή της ε, ελευθερίας διέλευσης που καθορίζεται στο άρθρο 5 του ΓΑΤ που επιτρέπει στα κοινοτικά σκάφη να εκφορτώνουν είτε για, ε, μετα ε, για εκφόρτωση είτε για τεκφόρτωση κάποια σημεία. Ο Επίτροπος ε, Μάντελσον από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου το 2000, συλλαμβάνοντας υπόψη και τις διαμαρτυρίες που είχαν γίνει για τα ε, σκάφη βαθέων υδάτων που ψάρευαν σε διεθνή ύδατα, επαναλαμβάνω διεθνή ύδατα, τα οποία ρυθμίζονται από τη ΣΥΕΤ, την Περιφερειακή Οργάνωση Αλληλεγγύας που είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Ο κύριος Μάντελσον λοιπόν τότε και θεώρησε και είχε απόλυτο δίκιο ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προσκόμματα κατά του ελεύθερου εμπορίου και γι' αυτό ακριβώς ε, προσέφυγε στην, στον Οργανισμό Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ. Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρξει μια αλληλοσυνεννόηση με τη Χιλή για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτή τη διαφορά και για να μπορέσουμε να αποσύρουμε την προσφυγή που είχε ξεκινήσει ε, στον ΠΟΕ. Πράγματι ήταν μια προσωρινή συμφωνία, πρόκειται για κάτι το οποίο μοιάζει πολύ με αυτό που έχουμε σήμερα και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες οι οποίες ήταν ε, εξελίξει εκείνη την εποχή. Ποια είναι τα δύο βασικά στοιχεία αυτού του μνημονίου. Καταρχάς υπήρχε ένα επιστημονικό πρωτόκολλο, ένα επιστημονικό πρωτόκολλο το οποίο τότε, επειδή αναφέρθηκε σας το λέω, το υπέγραψα διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναθέσει στην Ισπανία να κάνει την συμφωνία αυτή με τη Χιλή. Υπογράψαμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία την οποία σαφέστατα παραβίασε η χιλιανή πλευρά και γι' αυτό ακριβώς και διεκόπη. Και δεύτερον υπήρχε ένα σαφής στόχος που ήταν ο εξής δεδομένου ότι η Χιλή δεν ήταν συμβαλόμενο μέρα της περιφερειακής οργάνωσης αλληλείας που ρυθμίζει όλα αυτά τα ύδατα και θα σας εξηγήσω αργότερα για ποιο λόγο δεν είναι συμβαλόμενο μέρος η Χιλή. Συζητήθηκε αυτό διότι η Χιλή είπε θα ήθελε να κάνει μια διαφορετική ρύθμιση για την περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπεσε στην παγίδα και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Χιλή γιατί ήταν άλλο ένα από τα στοιχεία τα οποία ανέφερε το μνημείο. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο κ. Σπένσερ, ο οποίος τότε ήταν αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις για τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας δεν υπήρξε δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Χιλή ή να κάνουμε μια διαφορετική, διαφοροποιημένη περιφερειακή οργάνωση αλίας ή να δεχτεί η Χιλή να συμμετέχει στη ΣΥΑΤ. Πρέπει να πω ότι το ουσιαστικό πρόβλημα που υπάρχει στη Χιλή διότι εδώ προκύπτει αυτό το μνημόνιο το οποίο είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο. Στο προηγούμενο δεν τηρήθηκε τίποτα ούτε το επιστημονικό ε, πρωτόκολλο, αλλά ούτε και η δυνατότητα ε, πρόσβασης στους λιμένες. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Το 2004 υπήρξε διάταγμα από πλευράς χιλιανών αρχών, το 123 κάθετος 2004, στο οποίο και πάλι δημιουργούσαν προβλήματα για τη χρήση των λιμένων από τους κοινοτικούς στόλους. Και για να φτάσω στον ψηφία, διότι αυτό συζητάμε, προκύπτει το ίδιο πρόβλημα και για τον ηλιονδικό στόλο, ο οποίος ε, προσπαθεί να αλλιεύσει ε, για τα θέματα της ρέγκας. Εδώ υπάρχει άλλο διάταγμα του 2008 που έχει τα ίδια εμπόδια τα οποία τίθενται και για το ε, διάταγμα του 2004. Από πού προκύπτει όλο αυτό το πρόβλημα με τη χιλή προκύπτει από το γεγονό ότι η Χιλή δεν δέχεται οι περιφερειακές οργανώσεις αλληλεία σε μετανασταυτικά είδη να μπορούν να δίνουν συστάσεις που επηρεάζουν την οικονομική ε, ζώνη αλληλεία του. Επίσης, θέλει να μην επιτρέψει σε αυτούς που αλλιεύουν σε διεθνή ύδατα και θέλουν να βάλουν ε, τα δικά τους μέτρα ε, διατήρησης των αποθεμάτων και με όλα αυτά τα διατάγματα, διότι τα έχω διαβάσει όλα αναλυτικά, απαγορεύουν πρόσβαση στους λιμένες τους. Και εδώ υπάρχει λοιπόν σαφές πρόβλημα ε, παραβίασης διεθνούς δικαίου και δεν υπάρχει καμία συνεργασία από πλευρά Χιλής με τις περιφερειακές οργανώσεις Έχω κι άλλα όμως. Η Χιλή ως ε, παράκτιο κράτος κάποια στιγμή ξεκίνησε τη διαδικασία τροποποίησης του πώς το λέμε τώρα μια σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και από εκεί προέκυψε η συμφωνία για ε, τα ε, μεταναστευτικά είδη και η Χιλή ήθελε να επιβάλλει τα μέτρα διατήρησης των αποθεμάτων εκτός των ε, χωρικών της υδάτων. Και έτσι η Χιλή δεν υπέγραψε τη σύμβαση των ε, Ηνωμένων Εθνών για τα υψηλώς μεταναστευτικά είδη, διότι δεν ήθελε να κάνει καμία παραχώρηση. Είναι ένα άκρος εθνικιστικό κράτος και δεν θέλει να κάνει καμία παραχώρηση και καμία παραβίαση στην ε, ζώνη ε, αποκλειστική εκμετάλλευσή της. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια συμπεριφορά από πλευρά Χιλή η οποία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία. Η Χιλή εξακολουθεί να έχει τα δικά τη διατάγματα τα οποία επιβάλλουν σε διεθνή ύδατα συγκεκριμένα ε, κανόνες για να μπορούν να καθορίσουν τους δικούς τους κανόνες, ενώ η Χιλή εξακολουθεί να καταναλώνει και ξέρετε ότι υπάρχει μία διαδικασία νέας εθνικοποίησης. Ε, πέρα από τα χωρικά όδια, θα θέλουν να φτάνουν και να διευρύνουν τα ε, επιτρεπόμενα ε, μίλια και θέλουν να μην επιτρέπουν και στα σκάφη που έρχονται από την Ασία και τον Ειρηνικό να αλλιεύουν στις περιοχές τους και καταλαβαίνετε ότι με το προηγούμενο που έχουμε δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κάποιον ο οποίο παραβιάζει σαφέστατα όχι μόνο του κανόνε του ΓΚΑΤ αλλά και το δίκαιο της θάλασσα και διεθνεί κανόνε. Εγώ μίλησα με τον ε, ε, τομέα και μου λένε ότι προτιμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία η οποία καθορίζεται από τον ΠΟΕ και να μην υποκύψουν ε, στις απαιτήσει της Χιλής. Επειδή αυτό το μνημόνιο είναι το παλιό, το οποίο εδώ και 8 χρόνια δεν έχουν τηρήσει και επειδή η Χιλή ε, θεωρεί κάποια πράγματα όπως τις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας και τα ε, συμβάσεις υψηλώς μεταναστευτικών ειδών ως ε, άχρηστες, θα ήθελα να τηρήσουμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να περιμένουμε να λυθεί το θέμα ε, στον ΠΟΕ και να μην ε, υπογράψουμε κάτι το οποίο δεν θα τηρήσει κανείς όπως έγινε και στο παρελθόν. Δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα και θα ήθελα να καταψηφίσουμε την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα είναι δύσκολο να παρέμβω εγώ με την ίδια θέρμη. Δεν είναι βέβαια και πρόθεσή μου εδώ να προσπίσω τη χιλή, διότι πολλά από τα θέματα τα οποία ανέφερε η Πρόεδρος είναι ορθά ε, σε θέματα διεθνούς δικαίου. Και για τη συμπεριφορά της ε, χιλής, ε, κυρίως στις αρχές του 2000. Βέβαια, κάποια πράγματα εξελίσσονται και ευτυχώς κάποια πράγματα αλλάζουν. Η θέση της Χιλής ε, για την ε, Συμφωνία της Νέας Υόρκης δεν έχει αλλάξει βέβαια. Αλλά δεν είναι σωστό να λέμε ότι η Χιλή δεν έχει κάνει καμία πρόοδο για την στάση που έχει για τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις και τις πολυμερείς ε, οργανώσεις. Επί το πιο πρόσφατα παράδειγμα, στη νέα σύμβαση για το ε, νότιο ειρηνικό, για τα θηνοειδή, την υπέγραψε η Χιλή πολύ νωρίτερα από εμά, διότι εμείς θα ψηφίσουμε στις 26 Ιουλίου, ενώ η Χιλή την έχει ήδη ψηφίσει, ε, υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Είναι αλήθεια όμως ότι η Χιλή, στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης, η Χιλή παρουσίασε κάποιες θέσεις, σαν αυτές που μόλις μας περιέγραψε η Πρόεδρος, ε, επιμένοντας ότι θα πρέπει να υπερισχύουν τα εθνικά μέτρα, τα οποία κατά την άποψή τους θα έπρεπε να ισχύουν και στην ανοιχτή θάλασσα. Στη διάρκεια βέβαια αυτής της διαπραγμάτευσης η θέση τους άλλαξε και η οργάνωση αυτή θα λειτουργήσει ως περιφερειακή οργάνωση αλληλεία ε, συνήθης και η Χιλή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ε, διεθνείς οργανώσεις στο μέλλον, ακόμα και σε κάποιες οργανώσεις τις οποίες δεν ε, συμμετέχει αυτή τη στιγμή. Ένας από τους στόχους αυτής της συμφωνίας είναι ακριβώς να συνεχίσει η συνεργασία προκειμένου αν θέλετε να κοινωνικοποιηθεί η Χιλή και να αρχίσει να συμμετέχει σε αυτές τις διεθνείς οργανώσεις. Και αυτό ακριβώς συνέβη για τον Νότιο Ορεινικό, για την οργάνωση του Νοτιού Ορεινικού. Θα πρέπει βέβαια εδώ να πω ότι δεν είναι αλήθεια ότι αυτή η συμφωνία είναι πανομοιότυπη με αυτή του 2001. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκε βάσει της εντολής, όπως υπενθυμίστηκε, εντολή του Συμβουλίου, η οποία μας ζητούσε να διαπραγματευτούμε για να καθορίσουμε μία μόνιμη συμφωνία επί τη βάση της προσωρινής ε, συμφωνίας του 2001, η οποία ήταν ενισχύ. Δεν είναι αλήθεια ότι οι δύο συμφωνίες είναι πανομοιότυπες. υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ομοιάζουν, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα και γι' αυτό ακριβώ προτείναμε στο Συμβούλιο να υιοθετήσει την απόφαση για την εφαρμογή και την κύρωση αυτής της συμφωνίας. Και ποια είναι αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Η πρόσβαση στους λιμένες στη συμφωνία του 2001 διασφαλίζονταν, όπως πολύ σωστά υπενθυμίσετε, μόνο στα πλαίσια ενός προγράμματος επιστημονικής έρευνας, όπως αποκαλούνται. Τα σκάφη ήταν μόνο τέσσερα, μόνο τέσσερα ευρωπαϊκά σκάφη μπορούσαν να εκφορτώσουν και οι ποσότητες που μπορούσαν να εκφορτωθούν ήταν πολύ περιορισμένες. Αν θυμάμαι καλά ήταν μόνο 1.200 τόνοι. Επομένως μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην παρούσα συμφωνία το άνοιγμα τριών λιμένων που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που βρίσκουμε στον, στη συμφωνία για το... Ε, κράτο λιμένα. Έχουμε και κάποιε εξελίξει γιατί έχουμε και αλλαγέ σε διεθνέ επίπεδο για την πολιτική των λιμένων. Έχουμε τρεις λιμένες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλο τον κοινοτικό στέολο χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός στις ποσότητες που θα εκφορτώνονται. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο ε, δέχτηκε η Χιλή στη νέα συμφωνία ενώ δεν υπήρχε στην προηγούμενη και δέχτηκε να το συζητήσει μαζί μας ήταν να ξεχάσει αυτή την απέτηση που είχε να εφαρμόζει τα δικά της μέτρα. Εδώ ήταν για το ελάχιστο εθνικό μέγεθος ε, ξηφία ε, στα δικά μας τα αλλιεύματα τα οποία γίνονται σε διεθνή ύδατα, το οποίο ήταν ένα από τα ουσιαστικά σημεία τη Συμφωνία του 2000, γιατί ήταν ένα από τα σημεία που δεν δεχόμασταν εμείς τότε, να εφαρμόζονται εθνικά μέτρα εκτός ε, ε, χωρικών υδάτων. Αυτό δεν το δεχτήκαμε ποτέ για αλλιεύματα τα οποία ε, αλλιεύονταν στα διεθνή ύδατα. Και γι' αυτό ακριβώς ε, δέχτηκε και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει στον ΠΟΕ. Αυτό έχει διαγραφεί πλέον από τη Χιλή. Υπάρχει μια πολυδιάστατη συνιστόσα εδώ, η οποία δεν είναι ακριβώς το ίδιο βέβαια με τη συμμετοχή της Χιλής στην αρμόδια περιφαρική οργάνωση, αλλά ξεκινούμε πλέον με σαφή μνήμα προς το πολυδιάστατο επίπεδο. Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι δεν ε, ενεκρίθηκαν ένα μέτρο διαχείρισης του ψηφία στην Περιφερειακή Οργάνωση Αλίας ε, παρά τις συστάσεις μας το 2008 και το 2009 και εκεί δεν συμμετέχει η Χιλή. Υπάρχουν δηλαδή και άλλοι παράγοντες που δεν επιτρέπουν να γίνει και μεγάλη πρόοδο στην περιοχή. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να πούμε ότι εάν ο κλάδος θεωρεί ότι θέλει να ξαναπροσφύγει ε, στον ΠΟΕ, αυτό θα το εξετάσουμε, αλλά νομίζω ότι αλλάζει η θέση μας σε σχέση με το 2000. Καταρχάς υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στους λιμένες. Εμείς όμως, όπως επίσης αναφέρθηκε, εξακολουθούμε να μην είμαστε 100% βέβαιοι ότι η χιλή θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία και να είναι όλα τέλεια. Και εδώ λάβαμε και κάποιες μέρημνες. Η προσφυγή στον ΠΟΕ, η οποία αποσύρθηκε και ανέφερε, το ανέφερε και ο εισηγητές, μπορεί να ξανανοίξει αμέσως, νομίζω εντός δύο μηνών, και μπορούμε να προσθέσουμε και νέα στοιχεία, εάν φυσικά διαθέτουμε τέτοια στοιχεία, και η υπόθεση θα ανοίξει αυτομάτως τον ΠΟΕ εάν η Χιλή δεν εφαρμόσει σωστά όλα όσα έχουμε συμφωνήσει σε αυτή τη νέα συμφωνία. Έχουμε λοιπόν και μία ρήτρα διασφάλισης που μας επιτρέπει να προστατευτούμε στην περίπτωση κατά την οποία η Χιλή δεν θέλει να εφαρμόσει αυτό το οποίο έχουμε γράψει στη συμφωνία. Επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι πλέον έχουμε πρόσβαση στους λιμένες. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν ε, βάσει της ε, συμφωνίας ε, για το κράτος λιμένα, αυτά τα οποία έχουμε εγκρίνει και εμείς ε, στον κανονισμό για την παράνομη λαθρέα και αναρχελία για τις ε, τρίτες χώρες και τους λιμένες τους και φυσικά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί και εμείς και να τους δώσουμε ένα κάποιο περιθώριο δράσης ε, και εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, η οποία μας στήχησε και χρόνια δουλειάς και φυσικά επιτρέπει πλέον στο στόλο να εκφορτώνει ξηφία χωρίς προβλήματα στους τρεις λιμένες που έχουν δεθεί. Ξαναλέω βέβαια ότι εγώ δεν υπερασπίζομαι εδώ τη χιλή, απλώς προσπαθώ να υπερασπιστώ το θέμα της επίλυσης ε, του προβλήματος αυτού, το οποίο φυσικά είχαμε και την εντολή να επιλύσουμε. Από εκεί και πέρα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν. Ευχαριστώ επειδή και εγώ είμαι πρόεδρος, θα ήθελα να κάνω όλα προ ε, σχόλια. Ε, του. Why don't you take the... Κύριε Κάντεκ, θέλετε να αναλάβετε, γιατί εγώ θέλω να κάνω και άλλες ε, ερωτήσεις. Euh, ναι, ναι, Κάρμεν, κάνεις ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις, κανένα πρόβλημα. Ε, Κύριε Τσέζαρη, μας πήρε 20 χρόνια να ξαναβρεθούμε στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Δεύτερον, για την ορθή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας η ε, Χιλή θα πρέπει να παρεκκλίνει από μία σειρά από διατάγματα. Αν θέλετε μπορούμε να τα ζητήσουμε και αργότερα κατηδίαν γιατί δεν θα τα αναφέρω εδώ ένα-ένα. Αλλά ε, θα πρέπει να παραβιάσει και κάποια άρθρα του νόμου Αλίας που έχει η Χιλή. Εγώ επιμένω λοιπόν, εάν δεν παρεκκλίνει η Χιλή σε όλων αυτών των ε, θεμάτων που αναφέρονται στη συμφωνία το να υπογράψει τη σύμβαση για τα μεταναστευτικά, ήδη όταν ήταν οι πρώτοι που απέτησαν ε, να υπάρξει αυτή η συμφωνία θα είναι σαν να ζητάμε πολύ, Βέβαια το απαιτούμε από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω χιλή γιατί πρέπει να έχει ε, διαφορετική μεταχείριση. Αλλά όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς στη συμφωνία δεν συνάδουν με πάρα πολλά από τα στοιχεία που περιλαμβάνει στο νόμο της Αλίας της και σε πολλά διατάγματα τα οποία έχουν ε, υπογράψει εκάστοτε κυβερνήσεις της Χιλής. Αυτό μου δίνει για άλλη μια φορά την απόδειξη ότι μετά από 20 χρόνια που προσπαθούμε να επιλύσουμε φιλικώ ε, το θέμα τη διαφορά μα με τη Χιλή, δεν καταφέρνουμε να το επιλύσουμε. Και αυτή η συμφωνία δεν θα τηρηθεί, Σα το λέω εγώ, σα το υπογράφω και ο κλάδο το γνωρίζει και ξέρει ότι θα, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει του λιμένε, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί του λιμένε του Περού που δεν του βολεύουν και ο Περού και δυστυχώ θα γίνω και λίγο... Ε, θα μιλήσω και λίγο άσχημα εδώ, θα ξεβρακωθούμε στη χιλή και θα τους κάνουμε όλες τις απαιτήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα τα προσπαθούμε να τα κάνουμε για να τα καθησυχάσουμε με τη χιλή. Η χιλή είναι μια υπέροχη χώρα, χώρα με εξαίρεση την αλία. Με τους χιλιανούς μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα, εκτός από τη συζήτηση για τη θάλασσα και την αλληλεία. Εκεί αμέσως αλλάζει η στάση τους και αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Ο ε. Συγχαρητήρια κυρία Πρόεδρε. Καταπληκτικός ο λόγος σα Γνωρίζετε βέβαια τόσο καλά το ζήτημα αυτό που πραγματικά δεν μπορούμε παρά να σα πιστέψουμε. Νομίζω ότι γνωρίζετε τα πάντα όσον αφορά την αλληλεία για την χιλή. Πρέπει εγώ να πω βέβαια ότι δεν είναι ο δικός μου τομέας αυτός. Μια βασική ερώτηση. Έχει επικυρώσει η Χιλή το Άγκλος, δηλαδή το δίκαιο της θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών έχει επικυρώσει το δίκαιο αυτό η Χιλή. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη. Αν κατάλαβα καλά τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τους λόγους που προέκυψε η διένεξη αυτή ήταν ότι η Χιλή ήθελε ο κοινοτικό στόλος να αρχίσει να εφαρμόζει το ελάχιστο μέγεθος του ψηφία, ό,τι εφαρμοζόταν δηλαδή από την πλευρά της Χιλής. Ήθελε να επιβάλλουν και σε εμά το κοινοτικό στόλο το ίδιο πρότυπα. Κατάλαβα καλά ο κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα όσα είπαμε σήμερα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θεωρούμε ότι έχει κάνει καταπληκτικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο είπαμε απλώς ότι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και αν περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα του επόμενου μήνες, τα επόμενα χρόνια, ακόμα και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία θα συζητούμε τα ίδια πράγματα. Πρέπει λοιπόν αυτό το κοινοβούλιο και η δική μας επιτροπή να υπενθυμίσουν στις αρχές της Χιλής ότι πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες των διεθνών οργανισμών. Έχει κυβέρνηση η χώρα αυτή, έχουν αρχές. Νομίζω ότι δεν είναι δικός μας ρόλος να τους υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους διεθνείς κανονισμούς. Ακούστηκαν πολλέ απόψει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το άρθρο 5 τη ΓΑΤ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και ότι θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία αυτή και εγώ αυτό θα έλεγα, είναι σωστικά η μόνη σύσταση που μπορώ να κάνω. Και εγώ πρόσφατα ουσιαστικά ενημερώθηκα για το ζήτημα αυτό και αν μου είχατε θέσει ερωτήματα πριν από τρει μήνε, θα γνώριζα όσο γνωρίζει η κυρία Λόβεν. Μην θεωρεί πάντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο δεν ακούει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούμε τι λέτε, παρακολουθούμε την κατάσταση. Στα Ιρλανδικά λέμε ότι τα πράγματα προχωράνε βήμα προς βήμα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κινηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο, βαθμία, και πιστεύω ότι και η Επιτροπή μας θα πρέπει να εγκρίνει την προσέγγιση την οποία εκθέσαμε πριν από λίγο. Να κινηθούμε δηλαδή στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και στα πλαίσια της ΓΚΑΤ. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Χιλή με τη στάση της προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ουσιαστικά. Προσωπικά πιστεύω ότι εκφράζω και την άποψη των άλλων. Και βέβαια ακούστε τα όσα είπε η κυρία Φράγκα, η οποία είναι η δήμον στο ζήτημα αυτό. Να επιμείνω απλώ. στο γεγονό ότι έχουμε μια συνεννόηση η οποία διαφέρει από την προηγούμενη και απλώς θα πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε ε, πότε θα αποσύρουμε την προσφυγή στον ΠΟΕ, να έχουμε αφήσει να περάσει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, να διαπιστώσουμε ότι τηρούνται τα τη συμφωνία και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το κείμενο είναι το πλέον κατάλληλο και λογικό. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να μας εμποδίζει να ε, παραμείνουν τεχνητός οι διαφορές ε, και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μία συνεννόηση ε, και να έχουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Ο κύριος Τσέζαρη από την Επιτροπή. τα απάντηση, δεν αμφιβάλλω. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω δεν νομίζω ότι το κύρωσαν αυτό όπως και τη συμφωνία τη Νέα Υόρκη. Όσον αφορά τώρα τα εθνικά μέτρα, αυτά ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν τον κλάδο στην ε, ε, καταγγελία η οποία έφτασε μέχρι τον ΠΟΕΠ. Αυτό για τα ελάχιστα μεγέθη ήταν ένας από τους παράγοντες, αλλά πράγματι οι χιλιανοί να επιβάλλουν ε, το ελάχιστο αυτό μέγεθος το δικό τους ε, ε, στα είδη που αλλιεύουμε εμείς στα διεθνίδατα. Θα ήθελα απλώς να σας πω αγαπητοί ευρωβουλευτές ότι η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε στα πλαίσια της εντολής που της δόθηκε το αρχικό αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει άνοιγμα των λιμένων αυτών. Μπορούν να προσέλθουν τα σκάφη και να εκφορτώσουν. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να το περάσει η Χιλή στον ΠΟΕ. Δεν είμαι εγώ επιρρογνώμονα σε θέματα ΓΚΑΤ και ΠΟΕ, αλλά μέχρι τώρα υπήρχε ε, πρόβλημα στην πρόσβαση στους λιμένες. Επίσης δεν είμαι επιρρογνώμονα στην νομοθεσία της Χιλής, αλλά Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή θα έχουν υπογράψει μια διεθνή συμφωνία. Αυτή θα κυριαρχεί των ε, ε, χιλιανών διαταγμάτων που έρχονται σε αντίθεση με τα όσα έχουμε. Τώρα δεν ξέρω ποιο έκανε τη διαπραγμάτευση, αλλά φαντάζομαι ότι ο Χιλιανό που διαπραγματεύτηκε γνώριζε την προσωπική του νομοθεσία. Επομένω, φαντάζομαι ότι μάλλον ήξερε τι έκανε όταν διαπραγματευόταν. Τώρα, για το κατά πόσο θα γίνει σεβαστή ή όχι αυτή η συμφωνία, ειλικρινά αυτό νομίζω μόνο ο καιρό θα το δείξει. Αυτή τη στιγμή στεφτεί σε εφαρμογή η συμφωνία. Εγώ δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι έχουν υπογράψει μια συμφωνία με συγκεκριμένα στοιχεία δεν υπάρχουν εθνικά μέτρα τα οποία θα ισχύουν για τα λεύματά μας σε διεθνή ύδατα, δεν κλείνουν οι λιμένε. υπάρχει μια τεχνική και επιστημονική συνεργασία και υπάρχει μια πολυμερή συνεργασία. Αυτά τα βλέπετε στη συμφωνία, από εκεί και πέρα ε, μπορείτε να εξετάσετε το κείμενο και ε, να δείτε τι άλλο μπορείτε να δείτε. Κύριε Γκάλαχερ, θέλετε να πάρετε πάλι το λόγο μετά τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αρχική μου παρέμβαση και η τελική παρέμβασή μου ήταν νομίζω πολύ σαφής. Νομίζω ότι οι περισσότεροι στην Επιτροπή πιστεύουν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μέσω της ΓΚΑΤ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αποφανθούμε βέβαια σήμερα ή αν θα πρέπει να ψηφίσουμε κάποια άλλη μέρα. Εγώ πάντως προτείνω να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο μέσω της ΓΚΑΤ και στείλουμε ένα σαφές μήνυμα κατά αυτόν τον τρόπο προς τις αρχές της Χιλής. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκάλαχερ. Στις 30 Αυγούστου θα εξετάσουμε λοιπόν την έκθεση αυτή και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να πάρουμε και μια απόφαση. Πάντως, όπως το είπατε και εσείς κύριε Γκάλαχερ, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ στην αίθουσα που συμφωνούν με την προσέγγιση την οποία περιέγραψε η κυρία Φράγκα. Δεν είμαστε πάρα πολύ βέβαια στην αίθουσα, έχουν, στην αίθουσα έχουν μείνει καλύτεροι πάντως. Κυρία Λεβίν, θέλετε να πάρετε πάλι το λόγο. Δεν δόθηκε απάντηση στην ερώτησή μου. Αν έχει επικυρώσει η Χιλή την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Δίκαιο της Θάλασσας, τον Γιούγκλος. Ναι, το έχουν επικυρώσει, μάλιστα. Ευχαριστώ. Από όσο κατάλαβα, νομίζω ότι το επιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι κυρίως αλληλευτικού χαρακτήρα και, όσο, και όχι τόσο εμπορικού. Έχουμε και το Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Δεν είναι και αυτή μια εναλλακτική λύση. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σας δώσω άμεσα μια απάντηση. Πάντως νομίζω ότι έγινε μια καλή ανταλλαγή απόψεων για το ζήτημα αυτό. Καθένα είπε την άποψή του για τις ε, αλληλευτικές αυτές συμφωνίες. Και πάλι πιστεύω ότι οι περισσότεροι είμαστε κατά της συμφωνίας αυτής, αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ. Ακόμα και αν βέβαια ο κύριο Σάντσε ή κάποιοι άλλοι δεν συμφωνούν με την άποψη αυτή, πιστεύω ότι οι περισσότεροι πλειοψηφία, αν τι άλλο, στέθουσα αυτή, θα το δούμε βέβαια αυτό και αργότερα, θα χρειαστεί να ψηφίσουμε, πιστεύω ότι οι περισσότεροι είμαστε κατά αυτή τη αλληλευτική συμφωνία. Κάποια προσωπικά σχόλια τώρα. Πριν από λίγο, ο συνάδελφο Γκάλαχερ είπε ότι δεν ακούμε πάντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι δεν μας ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα. Μόλον ότι μερικέ φορέ προσπαθούμε να μιλήσουμε δυνατά. Α μα ακούει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συχνά δυνατόν. Δίνω και πάλι το λόγο στην α, καταπληκτική μα πρόεδρο. Eh, Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το σημείο τη ημερησία διάταξη. Το χρονοδιάγραμμα ούτω ή άλλως το εξήγησε ο συνάδελφο ο κ. Καντέκ. Και να περάσουμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 15, και πάλι είναι εισηγητή ο κ. Γκάλαγκερ, Συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Σύχνε, Λίχτενστάιν και νορβηγια χρηματοδοτικοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί 2009-2014 και εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλληλείας 2009-2014. Κύριε Γκάλαγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Πρόεδρε, εδώ πέρα μιλάμε λοιπόν για συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, Λίχτενσταν και Νορβηγίας. Ισχύει εδώ πέρα η συμφωνία που καλύπτει τις χώρες ΕΖΕΣ και συγκεκριμένα την χρηματοδότηση προς τις χώρες αυτές προκειμένου να εξαλειφθούν οι οικονομικές διαφορές που μπορεί να έχουν με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα πιο συγκεκριμένα για την Νορβηγία Υπάρχει ένα αποκλειστικό χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια. Χρησιμοποιείται λοιπόν το ταμείο αυτό προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προγράμματα για τις ε, κλιματικές αλλαγές, για την ε, διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη ε, του ανθρώπινου δυναμικού και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και κάποια νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στους χρηματοδοτικούς αυτούς μηχανισμούς. Από το 2009 λοιπόν, και μετά τα ποσά έρχονται στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσημε λοιπόν διαπραγματεύσει τη Ισλανδία, το Λίχτενστάιν και την Νορβηγία για την περίοδο 2009-2014 ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2008 και παράλληλα με τι διαπραγματεύσει αυτέ ξεκίνησαν και συνομιλίε για την επέκταση δύο διμερών πρωτοκόλων αλλιές με την Ισλανδία και την Νορβηγία. Επίσης υπάρχει και ένα πακέτο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, περίοδο 2009-2014, το οποίο και αυτό εγκρίθηκε. Μολονότι υπάρχει πολύ σημαντική αύξηση στο ταμείο αυτό και στη χρηματοδότηση και πρέπει να πούμε και ότι ε, η συμμετοχή της Ισλανδίας στο χρηματοδοτικό μηχανισμό παραμένει ίδια μολονότι υπάρχει έντονη οικονομική κρίση στη χώρα, όπως το γνωρίζετε. Πέρα λοιπόν από την συμφωνία αυτή χρηματοδότησης, ενονεώθηκαν δύο, τα δύο ελευτικά πρωτόκολλα. Θα δείτε στα παραρτήματα του εγγράφου ότι καταφέραμε να εγκρίνουμε τους μηχανισμούς αυτούς χρηματοδότησης προς την Ισλανδία και την Ορβηγία, αλλά και τα πρωτόκολλα, τα επιπλέον αλληλευτικά πρωτόκολλα. Καλύπτονται εδώ πέρα και οι χώρες ε, της πελαγικής ζώνης και της βόρειας ζώνης και ενδεχομένως υπήρχαν κάποιες ανησυχίες ότι ε, είχαν αυξηθεί οι ποσοστώσεις για συγκεκριμένα αλλιευτικά είδη. Αυτό δεν μας αφορά εμάς άμεσα στα πλαίσια της συμφωνίας, αλλά θεώρησα ότι θα πρέπει να το αναφέρω και αυτό, γιατί είχε προκύψει ως ανησυχία. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Εξ ονόματος Επιτροπής να δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Μέγερ από τη Ρελέξ και κατόπιν και μετά στον κύριο Ρόγκο Θαπατέρο από τη Γενική Διεύθυνση Κύριος... Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση, διότι ο κύριος Γκάλεγκερ αναφέρθηκε εις ε, ε, τα... Ε, τη συμφωνία για τα ψάρια τα οποία ελεύθησαν η ε, υπόψη. Ο κύριος Μέγερ πρώτα, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για την παρουσίαση της προτάσης, έχετε το λόγο. Thank you very much, Chair. Um... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκάλαγερ για την πολύ σωστή παρουσίαση που έκανε της κατάστασης. Θα ήθελα να πω πάρα πολύ σύντομα ότι μπορώ να δώσω ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία διότι ε, εφαρμόστηκε η, συμφωνία ε, για τις οικονομικές συνδρομές αλλά το 2004 με τη διεύρυνση ε, διαπραγματευτήκαμε δεκαπλή αύξηση σε αυτές τις ε, οικονομικές συνδρομές. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να εξετάσουμε το πρωτόκολλο της αλίας. Όταν τροποποιήθηκε το πρόγραμμα αυτό το 2007, όταν δηλαδή προσχώρησαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, στη περίπτωση αυτή, όπως εξηγήθηκε πάρα πολύ σωστά, λόγω της κατάσταση στην Ισλανδία πολύ σύντομα συμφωνήσαμε να αυξήσουμε τις συνδρομές αλλά α, θέλαμε να συμμετάσχουν και σε αυτή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γι' αυτό και ε, συνήφθη ένα πρωτόκολλο για την ε, Ισλανδία το οποίο ανανεώθηκε στα ίδια επίπεδα. Πρέπει να σας πω ότι καταφέραμε να έχουμε μία πολύ σημαντική ε, γενική αύξηση για την πενταετία και τα πρωτόκολλα αυτά τα οποία ανανεώθηκαν για την ίδια περίοδο περίχαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τρόπον ώστε να συμφωνήσουμε με την Νορβηγία στα πλαίσια του Συμβουλίου ότι θα προσθέταμε 250.000 τόνους γαρίδα και 350.000 τόνους ρέγγα. Ε, στα άλλα είδη δεν υπήρξε καμία αύξηση, μόνο αυτοί οι 250.000 τόνους για τη γαρίδα και 300 με 500.000 τόνους ρέγγα ε, που περιλαμβάνονται στη νέα αυτή συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτές ε, οι ποσότητες ε, που προσφέρονται στην Ισλανδία και στην Ορβηγία υπομορφής, υπομορφήν δασμολογικών ελαφρύνθεων δεν αυξήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό σε αυτή την τελευταία διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις δύο χώρες. Γι' αυτό το διπλό ε, στοιχείο που έχουμε αλληλείας και χρημάτων. Έγιναν κάποιες ε, ρυθμίσεις Αυτά, όπως έλεγε ο συνάδελφος, ξεκίνησαν το 2004 και πρέπει να πούμε ότι ανταποκρίνονται και σε μία ένδειξη καλής θελήσεως από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα επικοδομητικό πνεύμα, προκειμένου να αποζημιωθεί η Νορβηγία γιατί, ε, λόγω των επιπτώσεων της διεύρυνσης. Διότι πρέπει να πούμε ότι όταν η, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε με 10 χώρε αρχικέ, ε, στι οποίε προσετέθηκαν στη συνέχεια η Βουλγαρία και η ε, Ρουμανία. Κάποιε από αυτέ τι χώρε είχαν ε, ε δασμού δασμούς με την Νορβηγία και μετά με την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνετε ότι αυξήθηκε γι' αυτό ακριβώ και του προσφέρονται και αυτέ οι ελαφρύνσει, οι οποίες συνδέονται και με αυτή τη χρηματοδοτική συνεισφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιο το λόγο. Αν όχι, ολοκληρώθηκε και αυτό το σημείο και να πούμε το εξής. Η ανταλλαγή απόψεων Συγγνώμη, η παρουσίαση της νομοδότησης θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου. Ψηφίζουμε 26 και 27 Οκτωβρίου στην Επιτροπή. Κλείνουμε λοιπόν με το σημείο 15 και περνάμε στο σημείο 18 που αφορά τη Μεσόγειο και τα τεχνικά μέτρα για τη Μεσόγειο. Όπως γνωρίζετε, αποφασίστηκε η συνεδρία των συντονιστών να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει να μας εξηγήσει πώς ε, τίθενται σε πρακτική εφαρμογή αυτά τα μέτρα για τον περιβόητο κανονισμό των τεχνικών μέτρων της Μεσογείου. Οι τελευταίες παρακλήσεις αυτού του κανονισμού ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο φέτος και θα θέλαμε να ξέρουμε τι συνέβη με τα προγράμματα διαχείρισης, με την κατάσταση της ε, τήρησης των κανόνων και έχουμε καλέσει και την Περιφερειακή Οργάνωση της Μεσογείου. Έχουμε δύο προσώπους του ΡΑΚ, τον κύριο Φίλιο Μπαρναβάης και τον κύριο Μπονφίλιο. Καταρχάς λοιπόν και πριν δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο κύριο Δανατέλα είναι αυτός ο οποίο θα παρέμβει. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως, υπό μορφή εισαγωγή. θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσω την κατάσταση για την εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο και να εντοπίσω τις βασικές δυσκολίες τις οποίες έχουμε αναλύσει ότι αντιμετωπίζουμε και, και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των κρατών μελών και του τομέα διότι ο κανονισμός για την Μεσόγειο έχει οθετηθεί πριν από τρία χρόνια αλλά μόνο από λίγες εβδομάδες και συγκεκριμένα από τις 31 Μαΐου το σύνολο των διατάξεων έχουν όντως εφαρμοστεί. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι το βασικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εμείς θεωρούμε, όπως θεωρούσαμε ευθύς εξ αρχής, ότι πέραν των ε, προσωρινών αποκλήσεων που είχαν χορηγηθεί κατά την μεταβατική περίοδο ε, μέχρι τις 31 Μαΐου, οι περισσότερες διατάξεις όντως ε, εφαρμόζονταν. Οπότε πρέπει να θεωρήσουμε ότι η 31 Μαΐου είναι τελική ε, στάση στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιμένει αυτή την ημερομηνία για να αναλάβει ε, δράση στα θέματα των επιθεωρήσεων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού. Όπως ελέγχθη κανονισμό αυτό υπάρχουν ορισμένες πτυχές εκ των οποίων το πιο βασικό για, τη, για εμάς ε, προέρχεται από την λογική και την εφαρμογή του κανονισμού δηλαδή η υιοθέτηση των προγραμμάτων διαχείρισης management plan και πρέπει να σας πω ότι εν αντιθέσει με ό,τι αναφέρθηκε στο παρελθόν δεν είναι τα προγράμματα αυτά μόνο για να μπορεί κανείς να χορηγήσει εξαιρέσεις. Τα προγράμματα τα οποία προβλέπονται είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο για να επιτραπεί στα κράτη-μέλη και στους άμεσα εμπλεκομένους να υιοθετήσουν μέτρα και τεχνικές εφαρμογές κατά τρόπον ώστε οι διατάξεις του κανονισμού και οι πόροι να την χάνουν της καλύτερης δυνατής χρήσεως. Τα διαχειριστικά αυτά προγράμματα ε, έφτασαν πάρα πολύ αργά, άλλοτε ήταν ε, ε, ε, ε, ατελεί ή περιείχαν στοιχεία που δεν συνείδαν με τον κανονισμό και χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες πρέπει να σας πω ότι σήμερα για κανένα κράτος μέρος δεν υπάρχει σαφής κατάσταση ακριβής όσον αφορά τα διαχειριστικά προγράμματα. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα που έχει σχέση με τις εξαιρέσεις διότι εφόσον δεν υπήρχαν ε, ως επτοπλίστων ε, προγράμματα διαχείρισης τα οποία να σέβονται τις διατάξεις όταν πρέπει να λάβει επίσημες αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χορηγήσει εξαιρέσεις ε, δεν είναι δυνατό να το πράξει μέχρι σήμερα και πολλές αιτήσει αυτού του είδου έχουν αποπεμφθεί μέχρι ότου φτάσουν φάκελοι πολύ πιο αιτιολογημένοι και πολύ πιο πλήρεις. Ε, και πάλι δεν πιστεύω ότι η ιδέα εδώ είναι να υπησέλθουμε στη, στα μέτρα να κράτος μέλος αλλά η ανάλυση που κάναμε μας οδηγεί στο να πούμε ότι τα κείμενα έφθεσαν πολύ καθυστερημένα στις περισσότερες περιπτώσεις οι περισσότεροι δεν ε, συνάδουν με τους όρους που προβλέπουν ε, οι κανονισμοί και ξεκινήσαμε με τα κράτη-μέλη έναν διάλογο όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να καταφέρει να διευκρινίσει το τοπίο μετά από αυτή την πολύ σύντομη παρουσίαση θα ήθελα να σας πω ότι παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δεν είναι πλήρως αρνητικό διότι διαπιστώσαμε ότι η επιτάχυνση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι 31 ε, Μαΐου τελείωναν οι προσωρινές εξαιρέσεις και αυτό επέτρεψε και πρέπει να το τονίσουμε να συνειδητοποιήσουν οι εθνικές Αρχέ αρχές και όχι μόνον, αλλά και οι τοπικές αρχές και ε, πολλές φορές ε, η Επίτροπός μας και στο Κοινοβούλιο αυτό διαπιστώσαμε συζητήσεις ε, και ακούσαμε τοποθετήσεις από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που μας είπαν ότι η οδός που χρησιμοποιεί αυτός ο κανονισμός είναι σωστός και ευαισθητοποιεί τις τοπικού τους τοπικούς συμμετέχοντες και υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ίσως καθυστέρησε τρία χρόνια μετά από την εφαρμογή του κανονισμού και τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε και όπου επίζουμε θα μας επιτρέψει ε, να ξεκινήσουμε τώρα έναν ουσιαστικό διάλογο με όλους τους συμμετέχοντες ε, οι οποίοι εμπλέκονται στην εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο. Στη συνέχεια, αν το επιθυμείτε και αν υπάρχουν ε, ερωτήσεις μπορώ να σας πληροφορήσω για τις πρώτες επιθεωρήσεις τις οποίες κάναμε συστηματικά και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε αυτές τις επιθεωρήσεις και στο μέλλον, όχι μόνο για να φέρουμε σε δύσκολη θέση τις εθνικές αρχές, αλλά για να αντιληφθούμε ποια είναι τα προβλήματα που ε, ανακύπτουν ε, ε, στην πράξη και οι επιθεωρήσεις τις οποίες κάνουμε μαζί με τις εθνικές αρχές είναι όντως μέσα που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τη σωστή κατάσταση επιτόπου και ως εκ τούτου είναι βασικά στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων. Δεν ήθελα λοιπόν να κάνω ένα πλήρη απολογισμό της κατάστασης. Ο κανονισμός είναι περίπλοκος και πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουμε μαζί. Έχουμε δυσκολίες, αλλά είναι ένας κανονισμός ο οποίος επέτρεψε τους τελευταίους μήνες να ξυπνήσει κάπως τους εμπλεκομένους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να σταθμίσουμε σωστά το τι συμβαίνει επί τόπου. Ε, ε, και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε πιο συγκεκριμένα συγκεκριμένα ερωτήματα. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στους δύο προσώπου του ΡΑΚ. Σας παρακαλώ να ε, αποφασίστε μόνοι σας ποιος θα μιλήσει. Δεν ξέρω, ο κύριος Μπερναμπέη πρώτα και ο κύριος Μπομφούλιο στη συνέχεια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαστε πολύ σύντομοι. Μιλώ ως ε, προεδρεύων ε, του ΡΑΚ της Μεσογείου. Είμαι ένας επαγγελματίας ο οποίος δραστηριοποιείται πάνω από 25 χρόνια στον τομέα της αλίας και από το 1986 και τούδε συμμετέχω σε όλες τις συνεδριάσεις της ad hoc ομάδας της Μεσογείου, συμμετείχα και στις διπλωματικές διασκέψεις της Μεσογείου και συμμετείχα και στο σεμινάριο της Αγκώνα, το οποίο οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους πόρους της Μεσογείου, στην πρώτη συνεδρίαση επαγγελματιών όλου του αλληλευτικού τομέα της Μεσογείου στην Νάπολη το 1996. Επίσης συμμετείχα ως εμπειρογνώμων στις ε, γνωμοδοτήσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο και επιτρέψτε μου να σας πω και παρτίμος... Κυρίως τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ξεκινάμε από τη βάση ε, το ότι η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα, ναι μεν μικρότερη από άλλες θάλασσες, αλλά έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει παραδοσιακή κατανάλωση, παραδοσία παράδοση κατανάλωσης αλευμάτων, πολύ μεγάλη παράδοση οργανώσεων, πολύ στεναρών ε, των αλλιέων της και ταυτόχρονα ο αλλιευτικός κόσμος της Μεσογείου διαθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. πρέπει να γνωρίζουμε και την γνώμη και την αξιολόγηση των επαγγελματιών του τομέα. Δυστυχώς ε, δεν μπορώ να είμαι πολύ αισιόδοξο ούτε με τον κανονισμό του 94 τον 1626, ούτε με τις δυσκολίες που παρουσιάζει στην εφαρμογή του ο κανονισμός 1977 του 2006, στον οποίο δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη η άποψη των επαγγελματών του τομέα. Αυτά από πλευρά μου. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μπονφίλιο, ο οποίο είναι Γενικό Γραμματέα τη Περιφερειακή Οργάνωση Αλία και θα μπορέσει να σα ε, ε, περιγράψει πολύ καλύτερα τι αποφάσει του ΡΑΚ για τι τεχνικέ εφαρμογέ αυτού του κανονισμού διότι οι επαγγελματίες και όλοι όσοι διαστηριοποιούμεθα στον τομέα ζητάμε πάρα πολλές φορές αυτό που ακούμε στις Βρυξέλλες, ένα πραγματικό διάλογο με τον κλάδο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω διότι μας δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψή μας εδώ στην Επιτροπή Αλίας. Υπενθυμίστηκε ήδη από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο κανονισμός αυτός στην πραγματικότητα εγκρίθηκε ε, εδώ και πάνω από τρία χρόνια και θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι αυτός ο κανονισμός ε, υπέφερε πολύ κατά την εφαρμογή του, θα το θυμάστε εσείς κυρία Πρόεδρε, από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι την τελική έγκριση τον Νοέμβριο του 2006 χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια, τρία χρόνια μέσα στα οποία οι εκπρόσωποι του κλάδου είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο σε όλα τα κράτη-μέλη της Μεσογείου εξέφρασαν αρκετές επικρίσεις, ε, αμφισβήτησαν το κείμενο του κανονισμού σε διάφορα σημεία. Δεν θα ήθελα να επισέλθω εδώ σε λεπτομέρειες, αλλά από όλες αυτές τις επικρίσεις σε γενικές γραμμές, ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε σε δύο βασικά θέματα. Πρώτον, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές γνωμοδοτήσεις κατάλληλες, ε, οι οποίες να αναφέρονται και στις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου. Ο κανονισμός παρουσίασε και παρουσιάζει μία προσέγγιση ε, για την ε, πολιτική διατήρηση, ο οποίος θεωρούμε ότι είναι πιο ε, κατάλληλος για τις ε, υπόλοιπες ευρωπαϊκές θάλασσες ε, και δεν λαμβάνει υπόψη στην αλληλεία πολλαπλών ειδών, ε, άνα συγκεκριμένο είδος, ε, άνα είδη τα οποία έχουν πιο μεγάλο κύκλο ζωής. Να υπενθυμίσω στη Μεσόγειο ότι είναι πολύ πιο μικρός ο κύκλος ζωής των αλευμάτων στη Μεσόγειο και αναφερόμαστε και σε μαζικά αλεύματα, ενώ στη Μεσόγειο είναι πιο διάσπαρτα και πιο διαφοροποιημένα τα είδη που αλεύονται. Ο βασικός κανονισμός λοιπόν, ο 1977, ε, βασίστηκε σε αυτά την έννοια. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε κανένα κράτος μέλος δεν μπόρεσε ακόμα να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα διαχείρισης το οποίο θα καταποκρίνει τις απαιτήσει του βασικού κανονισμού. Δεν είναι τυχαίο διότι δεν θεωρώ ότι κανένα από τα 7 μεσογειακά κράτη-μέλη έχει τεχνικές δυσκολίες. Υπάρχει προφανώς κάτι το οποίο δεν πάει καλά. Η δεύτερη ομάδα επικρίσεων αφορούσε το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία αξιολόγηση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων ε, αυτού του κανονισμού. Πράγματι, μέχρι τούδε κανείς δεν γνωρίζει σαφώς Πού πήγαν όλοι αυτοί οι αλληλείς οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τον κλάδο. Κανένας δεν ξέρει πού θα καταλήξουν όλοι οι αλληλείς οι οποίοι θα φύγουν στο μέλλον από τον κλάδο. Ε, όχι μόνο γιατί μειώνεται ο, στέλος, ε, ο στόλος, αλλά και γιατί ε, τέθηκε σε ισχύ αυτός ο κανονισμός. Από τον Νοέμβριο του 2006, ε, από τότε που εγκρίθηκε ο κανονισμός μέχρι τις 31 Μαΐου του 2010, δηλαδή πριν από λίγες εβδομάδες, υπήρξε περιορισμένη εφαρμογή του κανονισμού ε, χάρη στην ε, παράταση των ε, κάποιων κανόνων. Αλλά μόλις λήξει αυτή η παρέκκληση, την 1η Ιουνίου του 2010 δηλαδή, που έληξαν, άρχισαν και πάλι να ισχύουν αυτές οι επικρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, Ισχύουν οι κανόνες πλέον για το ελάχιστο μέγεθος ε, για το ε, παρασυρώμενο δίκτυ αλλά και για την απόσταση από την ακτή, όχι μόνο για το παρασυρώμενο δίκτυ και αναφέρονται κάποια στοιχεία γενικού χαρακτήρα για την διατήρηση των αποθεμάτων και θεωρούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι υπερβολικά για κάποιες περιοχές και για κάποια συγκεκριμένα ε, αλλιευτικά αποθέματα τα οποία μπορεί να είναι περιθωριακά για την αλληλεία εν γέννη, αλλά είναι πολύ σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες και για τις εποχιακές ε, αλληλείας. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες, ε, κατά 50% και αυτό φυσικά, επειδή ακριβώς η μείωση είναι στο 50%, θα υποχρεωθούν πολλές επιχειρήσεις να ε, κλείσουν και θα ε, έχουμε και αύξηση του ποσοστού παρανομίας. Για την Βόρεια Δυραδική Σάλασσα ε, και τα παρασυρώμενα δίκτυα εκεί θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι αλλιεύονται ήδη μικρού μεγέθους τα οποία είναι ήδη ενήλικα. Γι' αυτό ακριβώς το ΡΑΚ τη Μεσοχείου που συνεδρίασε στις αρχές ε, Ιουνίου στην Ισπανία ετοίμασε μια επιστολή η οποία απεστάλλει στην Επίτροπο Δαμανάκη την οποία νομίζω ότι λάβανε και τα μέλη της επιτροπή σα και μέσω αυτής της επιστολής ζητούμε να μην υπάρχουν απλώς παρατάσεις και παρεκκλήσει, αλλά να γίνει μια κατεπίγουσα επαλήθευση που θα ε, επιταχύνει την αναθεώρηση που προβλέπει ο ίδιος ο κανονισμός το 2012. Ε, μία κατεπίγουσα επαλήθευση η οποία θα αξιολογήσει τους πόρους και τις δυνατότητες που έχουμε για να κάνουμε μία τροποποίηση τουλάχιστον για τις πιο προβληματικές πτυχές. Να υπενθυμίσω το θέμα του μέγιστου ε, μήκους του δικτύου που είναι πρόβλημα κυρίως ε, στην Ισπανία το ελάχιστο μέγεθος δικτύου που δεν επιτρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να αλλιεύονται κάποια ενήλικα είδη μικρού μεγέθους την ελάχιστη απόσταση από την ακτή σε κάποιες περιοχές και τη συνοχή όλων αυτών με τα ελάχιστα μεγέθη. Επιπλέον, κυρία Πρόεδρε, και θα πρέπει εδώ να το υπενθυμίσουμε αυτό, στη Μεσόγειο η πολιτική διατήρηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει μόνο για την βόρειο-ανατολική πλευρά της λεκάνης της Μεσογείου και στις άλλες περιοχές αρχίζει να αυξάνεται η αλία παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένε συστάσεις του ε, Γενικού Συμβουλίου Αλίας της Μεσογείου και έχουμε ένα συνολικό ποσοστό το οποίο αποζημιώνει ουσιαστικά τη μείωση της ευρωπαϊκής αλλιευτικής δυνατότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό το θέμα της διαχείρισης των αποθεμάτων της Μεσογείου και δεν είναι κατανοητό και εύκολα αποδεκτό το γεγονός ότι περιορίζεται, ε, κάποια, περιορίζονται κάποια στοιχεία από την κοινή αλληλευτική πολιτική και έτσι οι αλληλείς μας είναι λίγο εχθρικοί προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί οι όροι όπως η εναρμόνιση των τεχνικών μέτρων διαχείρισης της λεκάνη στη Μεσογείου, ανα διάρθρωση ή διαφοροποίηση των αλλιευτικών δυνατοτήτων εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και αυτοί οι όροι προς το παρόν ισχύουν μόνο επί χάρτου και δεν έχουν υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ανδρέας Μπαρέα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια επί του θέματος, διότι Οι σοσιαλιστές ε, ανεφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Αυτός ο κανονισμός για τα τεχνικά μέτρα είναι ένας δύσκολος κανονισμός, ο οποίος είναι καθόλου τεχνικός, ε, εγκρίθηκε πριν από τρία χρόνια και υπήρξε και διαβούλευση από το Συμβούλιο, αλλά έχουν ήδη περάσει τρία χρόνια και ήγηκε η ώρα να αξιολογήσουμε τις ε, δυσκολίες της εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα εφαρμογής που θα μπορούσαν να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος ε, του ΡΑΚ από την Ιταλία, ο οποίος μόλις ε, ολοκληρώσε την παρέμβασή του, το μέγεθος του ματιού, το μήκος του δικτυού, που δεν είναι μόνο θέμα προστασίας, αλλά το γεγονός ότι τα δίχτυα τα ίδια καταστρέφουν τα αλλιεύματα και μετά δεν μπορούν να απολυθούν και φυσικά ε, η απόσταση από την ακτή. Εγώ, κυρία Φράγα, δεν είμαι η δήμον του θέματος. Ε, φαντάζομαι ότι όσοι μίλησαν μόλις ε, σας τα εξήγησαν. Μας το λένε λοιπόν οι εκπρόσωποι του κλάδου. Αυτό το οποίο σαφώς ισχύει είναι το γεγονός ότι δεν ε, υπολογίσαμε και τις αποστάσεις ε, εις βάθος που ορισμένες φορές δημιουργούν προβλήματα στην αλία. Η θέση μας είναι ότι δεν είμαστε μεν κατά του κανονισμού, αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένε τεχνικές διευκρινήσεις και τεχνικές τροποποίησεις, ότι πρέπει να συμμετέχει ο κλάδος και ότι μιλάμε για ε, αλληλεία η οποία γίνεται πολύ κοντά ε, στις ακτές και υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Η Μεσόγειος θάλασσα είναι πάρα πολύ σημαντική ε, όπως και οι άλλες θάλασσες φυσικά, αλλά έχει κάποιες βασικές ανάγκες επιβίωσης, στοιχειώδεις ανάγκες, διότι ε, μία σειρά από χώρε οι οποίες όμως δεν τηρούν τους ίδιους κανόνες με εμά. Ξέρουμε ότι στη Βόρεια Αφρική δεν ισχύουν οι κανόνες, ε, ούτε βέβαια και στην, ε, στις άλλες χώρες. Μόλις μιλήσαμε για την Ισλανδία, αλλά στο Νότο ε, είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν μία αξιολόγηση αδικτύπου που από τεχνική πλευρά να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να γίνουν συγκεκριμένε τροποποίησεις και να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θα σας απαντήσω, διότι εγώ ήμουν εισηγήτρια επί του θέματος και το ξέρω πολύ καλά. Η κυρία Λεβί. Uh, okay, thank you. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι μου φαίνεται περίεργο ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον επαγγελματικό κλάδο τώρα. Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2006. Συνεπώς υπήρχε εξαίρεση από την εφαρμογή του κανονισμού αυτού για περισσότερα από τρία χρόνια και νομίζω τα κράτη-μέλη και ο επαγγελματικό κλάδο είχαν πάρα πολύ χρόνο για να αντιδράσουν. Όντως συμφωνήσαμε στην συνάντηση των στονιστών να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας μιλήσει για τα κράτη-μέλη αυτά που είχαν ζητήσει επιπλέον εξαίρεση από την εφαρμογή του κανονισμού. Δηλαδή, αίτηση που έγινε στις 31 Μαΐου. Δεν νομίζω όμως ότι συμφωνήσαμε στην συνάντηση των συντονιστών, στην ευρία των συντονιστών, έχουμε και άλλους προσκεκλημένους πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα δηλαδή ότι θα είχαμε εκπροσώπους του επαγγελματικού κλάδου, Ενδεχομένω στην περίπτωση αυτή να έπρεπε να είχαμε και κάποιου εμπειρογνώμονε, οι οποίοι θα μα εξηγούσαν για ποιο λόγο καταρτίζονται κατά αυτόν τον τρόπο τα προγράμματα διαχείριση. Θα μπορούσαν να απαντήσουν στην περίπτωση αυτή οι εμπειρογνώμονε στι επικρίσει που ακούστηκαν μόλι τώρα από τον ε, επαγγελματικό κλάδο. Ακούσαμε πάντω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 10 Μαου έστειλε μια επιστολή με υπογραφή του κ. Μοντέση προ το Ιταλικό Υπουργείο, αποδεχόμενη την ε, αίτηση εξαίρεσης της Ιταλίας για συγκεκριμένους τομείς, εξαίρεση από τον κανονισμό. Αληθεύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ εκνευρίζομαι. Ίσως δεν καταλαβαίνω, δεν κατανοώ το πρόβλημα και έχω δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν ε, κατάλαβα καλά το θέμα για το λίγο χρόνο που είμαι σε αυτή την Επιτροπή, οι ε, κανονισμοί συναποφασίζονται από το Συμβούλιο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλες οι κυβερνήσεις της Μεσογείου χρειάστηκε να συνενέσουν σε αυτόν τον κανονισμό. Δηλαδή θεώρησαν ότι ήταν ε, μία σωστή ρύθμιση. Έχω δίκιο. Δεύτερο ερώτημα. Εδώ υπάρχει μία μεγάλη επίπληξη και λέγεται ότι δεν υπάρχει επιστημονική παρακολούθηση και επιστημονικά στοιχεία ότι δεν υπήρξε συλλογή αυτών των στοιχείων που να χρησιμοποιηθούν για αυτό το νομοθέτημα. Θα ήθελα λοιπόν ευχαρίστως να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποια μορφή συνέλεξε τα επιστημονικά στοιχεία και βάσει ποιων ε, στοιχείων κατερτίστηκε αυτό το νομοθέτημα ήθελα να παρέμβω κι εγώ γιατί ήμουν εισηγήτρια επί του θέματος και θα ήθελα να γνωρίζετε κι εσείς πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το θέμα. Ο κανονισμός αυτός ο οποίος τροποποιούσε το προηγούμενο κανονισμό που επρόκειται για ένα κανονισμό εντελώς παροχημένο διότι όπως ε, θα σας επιβεβαιώσω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκριθεί σε ένα συμβούλιο με πάρα πολλές πολιτικές επιρροές ε, και τεχνικές ελλείψεις. Ήταν ένας τελείως αντιφατικός κανονισμός. Ε, ούτε καν το μέγεθος του ματιού δεν υπάκουε στα ελάχιστα μεγέθη, ήταν αδύνατον να τηρηθεί αυτός ο κανονισμός. Επειδή ακριβώ λοιπόν υπήρχε αυτή η αδυναμία, δεν τηρούνταν ο κανονισμό και δεν λειτουργούσε ο κανονισμό. Όπω ήταν λογικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα πρόταση που τροποποιούσε αυτόν τον κανονισμό, ο οποίο ήταν παντελώ άχρηστο, διότι δεν μπορούσε να τον τηρήσει κανεί. Και είχαμε μια πρόταση, η οποία ναι μεν είχε τα προβλήματά της, ε, την οποία σαφώς ο κλάδος απέρριψε και το Κοινοβούλιο σε πρώτη συζήτηση με τότε έναν Ιταλό εισηγητή από την πολιτική μου ομάδα, ο οποίος ε, γνώριζε καλά το θέμα, Χρειάστηκε να ξαναντιδράσει και να κάνει μια έκθεση, δόθηκε νέα εντολή και εγώ ανέλαβα από εκεί και πέρα την έκθεση αυτή, διότι γνώριζα φυσικά καλά τη Μεσόγειο, προφανές αυτό. Για πρώτη φορά λοιπόν και πριν ακόμα φτάσουμε σε αυτή την περιβόητη συναπόφαση, ε, διότι εγώ δέχτηκα να αναλάβω το θέμα αυτό με μόνη προπόθεση ότι ο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό που θα τροποποιούσε την πρόταση και έγινε παραδεχόμενη πάρα πολλά από τα αιτήματα του κλάδου τότε. Ε, προφανώς δεν μπορούσαμε να τα εγκρίνουμε όλα, διαγράψαμε όλα τα σημεία τα οποία ίσω δεν είχαν επαρκή επιστημονική υποστήριξη. Τέλο πάντων καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό που άλλαζε την πρόταση, μετά το Συμβούλιο άλλαξε κάποιο πράγμα μεταξύ αυτών άλλαξαν πολλά πράγματα για τι προτάσει για το ψηφία, για τα ε, νέα μήκη τα οποία ήταν απαράδεκτα και έγινε σεβαστό το οποίο εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω το άρθρο 13 που είναι η απόσταση από την ακτή που αυτή τη στιγμή αμφισβητείται και έγινε σεβαστό από απολύτως με μία και μόνη εξαίρεση που ήταν η ρύθμιση για του, α, υδραυλικά ε, τμήματα και έγιναν αποδεκτά όλα τα υπόλοιπα ε, και υπήρχε δυνατότητα τα κράτη-μέλη μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης να θέσουν εξαιρέσεις ακριβώς για τους λόγους στους οποίους περιέγραψε η κυρία Ανδρέας Παρέα. Ένα άλλο πρόβλημα βέβαια το οποίο προέκυψε είναι ότι τα κράτη-μέλη ή δεν το έκαναν ή δεν το δικαιολόγησαν. Και εδώ λοιπόν υπάρχει και μεγάλη ευθύνη των κρατών μελών που πλήττονται από αυτόν τον κανονισμό. Ε, επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό δεν έγινε και μόλις το επιβεβαίωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν έγινε είναι ε, υπέτεια τα κράτη-μέλη τα οποία δεν το αιτιολόγησαν. Ε, θεωρώ ότι έγιναν σεβαστά πολλά σημεία. Το θέμα είναι ότι στο κανονισμό αυτό προσαρμόστηκαν πολλά από τα ελάχιστα μεγέθη. Ε, θα θυμάστε το θέμα της Αρδέλας, ε, έγινε μια πρόταση που ήταν αντίστοιχη με αυτή του Ατλαντικού. Καταφέραμε να μειώσουμε το ελάχιστο ε, μέγεθος γιατί μας φάνηκε ότι ήταν πιο κατάλληλο το μέγεθος αυτό. Θέλω δηλαδή να πω ότι συζητήθηκε το θέμα με τον κλάδο και ο κλάδος λίγο πολύ δέχτηκε αυτή την πρόταση της οποίας την οποία είχαν συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και ήταν σαφώ καλύτερη από την αρχική. Αυτό που με εκπλήσει λοιπόν είναι που αντέδρασε τώρα ο κλάδο μετά από τόσα χρόνια και εξακολουθεί να μην τηρεί τον κανονισμό και τα κράτη-μέλη δεν παρουσιάζουν προγράμματα διαχείριση. Το θέμα είναι τι λύση μπορούμε να δώσουμε στο θέμα αυτό, διότι δεν νομίζω ότι η λύση είναι να ξαναρχίσει η συζήτηση για τον κανονισμό, για να ξαναθέσουμε όλα εκ νέου και να μην έχουμε τίποτα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και γιατί τα κράτη-μέλη δεν παρουσίασαν προγράμματα διαχείριση και γιατί εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η κατάσταση. Και εγώ θα ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι μέλη γενέστε, ποιο είναι το επόμενο βήμα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κανονισμό που δεν τηρείται. Ή χρησιμεύει ή δεν χρησιμεύει, ή κάνουμε εξαιρέσει ή τηρούμε τον κανονισμό. Ο κλάδο, τα κράτη-μέλη κάνουν τη δουλειά του ή δεν την κάνουν. Εγώ θα ήθελα να ξέρω όμως τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει την κατάσταση στη Μεσόγειο. Διότι το να έχουμε ένα νέο κανονισμό, καλό, κακό, καλύτερο, χειρότερο, ούτως ή άλλως είναι άχρηστο, διότι δεν τηρείται. Και θα ήθελα να επικρίνω τον κλάδο και δεν με πειράζει, διότι ούτως ή άλλως εγώ λέω τα πράγματα στα ράτα και με το όνομά τους. Ε, καλέσαμε εδώ το ΡΑΚ Μεσογείου, διότι θεώρησα ότι η Περιφερειακή Οργάνωση Αλία στη Μεσογείο μπορούσε να είναι παρούσα εδώ και αναλαμβάνω και την ευθύνη, εγώ τους κάλεψα, δεν το ζήτησαν αυτοί, εγώ δική μου πρωτοβουλία ήταν να του ζητήσω να είναι εδώ, διότι θα ήθελα να ακούσω την άποψη του κλάδου. Αν δεν συμφωνείτε, εγώ αναλαμβάνω πλήρω την ευθύνη. Αλλά μπορώ να κάνω μια επίκριση εδώ και να πω ότι η Περιφερειακή Οργάνωση Αλία τη Μεσογεία θα μπορούσε να είχε αντιδράσει νωρίτερα. Αφού δεν αντέδρασαν λοιπόν και περίμεναν να φτάσει η τελευταία στιγμή για να έχει τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμό και να έχουν λήξει οι τελευταίε εξαιρήσει, ε, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι. Ίσως θα μπορούσαν να είχαν βελτιωθεί κάποια πράγματα, τα θέματα του μεγέθους, να είχαν γίνει κάποιες μελέτες που να δικαιολογούσαν κάποια πράγματα, να είχαν γίνει κάποιες τροποποίησεις, οι οποίες όμως δεν έγιναν γιατί ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε ο κλάδος, ούτε κανείς δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να ισχύει ο κανονισμός. Και μου φαίνεται ότι είναι κρίμα το γεγονός ότι δαπανήθηκε τόσο χρόνο και σα το λέω εγώ γιατί εγώ εργάστηκα για την έκθεση, συνεργάστηκα με την Επιτροπή. Εμείς στο Κοινοβούλιο το πήραμε πολύ στα σοβαρά το θέμα και διαπιστώσαμε διαπιστώνω ότι η κατάσταση είναι ίδια. Και λέω και κάτι ακόμα και μετά θα σταματήσω. Το γεγονός ότι δεν τηρούνται κάποια πράγματα στη Μεσόγειο, δεν τηρούνται τους κανόνες στην Αλία, στη Μεσόγειο, δεν ε, ε, έχει σχέση απλώς με το γεγονός ότι έχουμε ένα κανονισμό που ίσως θεωρείται ότι δεν είναι κατάλληλος για τη Μεσόγειο το επειδή δεν τον τηρεί κάποιο τον κανονισμό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εμεί κανονισμού και να μην του τηρούμε, διότι εμεί είμαστε αυτοί οι οποίοι αλλιεύουμε περισσότερο στη Μεσόγειο. Δεν μου αρκεί εμένα αυτή η η αιτιολογία ότι έχουμε και άλλες χώρες που δεν τα τηρούν αυτά τα πράγματα. Έχουμε κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να ισχύουν για όλους όπως τα μέτρα του ΓΚΑΤ κλπ. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι αιτιολογείται σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι επειδή στην Τινησία ας πούμε δεν τηρούν τους κανόνες πρέπει να μην τους τηράμε κι εμείς. Ε, πρέπει να τα παραδεχτούμε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν σχέση τα μέτρα που έχετε εσείς με τα μέτρα που έχουν στον Ατλαντικό γιατί και πάλι δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση. Μισό λεπτό ολοκληρώνω κυρία Ανδρέας Παρέα. Το ξέχασα το όνομά σα τι να σα πω, είμαι συγχυσμένη όλη μέρα εδώ στη συνεδρίαση. Εύκολο είναι, αλλά δεν σα βλέπω και πολύ συγχυσμένη, κυρία Φράγκα, λέει κυρία Ανδρέα Μπαρέα. εγώ νομίζω θα προσπιζόμουν με τον ίδιο τρόπο τα συμφέροντα τη ε, Μεσογείου, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ε, ότι δεν είναι ευθύνη μόνο των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη δεν αντέδρασαν με δικά τους προγράμματα διαχείρισης, ε, γιατί αφήσαμε να παρασυρθούμε με τα τρία χρόνια των εξαιρέσεων ε, της εφαρμογής του κανονισμού. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε. Δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το σύνολο του κανονισμού, διότι και πάλι άλλα δύο χρόνια θα δαπανίσουμε για να το κάνουμε, αλλά πρόκειται για ένα κανονισμό ο οποίος είναι πάρα πολύ τεχνικό και δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να τροποποιήσουμε όλα τα πράγματα. Θα πρέπει όμως να ξεκινήσει μία περίοδος περισυλλογής μετά από αυτά τα τρία χρόνια. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα και δεν είναι κανείς κατά του κανονισμού. Είμαστε κατά του γεγονότος ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και αυτό που θα θέλαμε εμείς είναι να έχουμε κανονισμό που να εφαρμόζεται. Εάν όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι κάποιος αλλιεύει στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή και αυτό που ε, ψαρεύεται πρέπει να πεταχτεί γιατί δεν ε, πουλιέται στο εμπόριο λόγω του μεγέθους του δικτυού, καταλαβαίνετε ότι δεν θα τηρείται ο κανονισμός. Και αφού δεν θα τηρείται ο κανονισμός πρέπει να τον αθεωρήσουμε να δούμε τι προβλήματα προβλήματα υπάρχουν, διότι είναι τεχνικά θέματα που έχουν λύση. Η κυρία Ρόντους. Λοιπόν, ε, ε ξέρω ότι θίγω τους μεσογειακούς συναδέλφους αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, εάν τελειώνουν οι μεταβατικές περίοδοι και, περίοδοι και αρχίζουμε να αμφισβητούμε τα θέματα, ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να εφαρμόσουμε ε, μεταβατική περίοδο. Είχαμε τρία χρόνια. Μπορούσαμε να έχουμε χρησιμοποιήσει την περίοδο αυτό να λύσουμε τα προβλήματα. Αν υπάρχουν όμως τώρα προβλήματα θα ήθελα να μου απαντήσετε στα ερωτήματα. Υπήρχαν, υπήρχαν επιστημονικά στοιχεία, συζητήθηκαν λύσεις πριν από την τον ομόφωνο κανονισμό του Συμβουλίου που υπερψηφίστηκε και αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα και εάν μας τα μετακυλά ε, το Συμβούλιο αναρωτιέμαι ε, πόσο τολμάει το Συμβούλιο να μας μειώνει τις πιστώσεις, πράγμα το οποίο συζητήσαμε πριν από λίγο, διότι δεν μπορεί να γίνει πλέον έλεγχος γιατί δεν έχουμε χρήματα ε, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάμε για το μέλλον της Ελίας υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας παρακαλώ, η Ντονατέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι δύσκολο να απαντήσω τώρα σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που όντως αποδεικνύουν ότι είμαστε σε μία φάση συγχρόνως αρχής ε, υλοποιήσεως του κανονισμού ο παρόλο που έχει οθετηθεί εδώ και τρία χρόνια όπως σωστά υπενθυμίσατε και αντιμετωπίζουμε προτάσεις, συστάσεις, συζητήσεις που ε, απαιτεί ο, κλάδος και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό σήμερα είναι απαραίτητο διότι υπάρχει μία ε, ανησυχία και πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η ανησυχία αυτή οφείλεται στην Επιτροπή διότι έχουμε ε, λήψεις πληροφοριών περιμένουμε να λάβουμε από τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία θα θέλαμε να έχουμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πραγματικά τον κανονισμό επιτόπου. Υπάρχει μία ανησυχία από τον κλάδο και δεν πρέπει εμείς να κρίνουμε αν οφείλεται στην ε, ε, αναμονή τριών ετών ή κάτι άλλο. Είναι κάτι όμως στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούμε. Και δεν είναι μόνο θέμα του ΡΑΚ αλλά και όλων των άλλων συμμετεχόντων όπου όλοι πρέπει να διευκρινίσουν σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Και υπάρχει και μια άλλη δυσκολία όσον αφορά τις εθνικές διοικήσεις για να μπορέσουν σήμερα να αντιμετωπίσουν έστω και καθυστερημένα καταστάσεις οι οποίες είναι περίπλοκες. Λοιπόν, όταν ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία απογραφή της κατάστασης του κανονισμού για τη Μεσόγειο, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση δεν μπορούσα να έρθω εδώ και να αναφερθώ για το σύνολο των χωρών και το σύνολο των περιοχών αναχώρα όλα τα διαχειριστικά προγράμματα που έχουμε εφαρμόσει, διότι έχουμε εκπονήσει χιλιόμετρα εγγράφων, έχουμε πίνακες που αντικατοπτρίζουν όλες αυτές τις πληροφορίες και είναι στη διάθεση όλων επιθυμούν ε, να γίνει μία πιο λεπτομερής και πλήρης παρουσίαση. Παίρνω σαν παράδειγμα ε, τα προβλήματα τα οποία έθιξε η κυρία Λεβίν, παραδείγματο χάρη. Αν στείλαμε επιστολές στην Ιταλία λέγοντας ότι δεχόμαστε ορισμένες προτάσεις, η απάντηση ήταν ναι, βεβαίως. Αλλά στείλαμε την ίδια επιστολή στην Κύπρο, στην Ισπανία, διότι υπάρξουν διατάξεις δεν είναι το ε, άρθρο 13.5 αλλά 13.11 του κανονισμού σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη ε, ε, πρέπει να υιοθετήσουν συγκεκριμένες διατάσεις για να εξαιρεθούν από την αλληλεία σε μία απόσταση από την ακτή με ορισμένους περιορισμούς. Και το διευκρινίζω σήμερα όχι γιατί έχουμε κάτι να κρύψουμε ή θέλουμε να αποφύγουμε τη συζήτηση, αλλά διότι αν θέλουμε να ασχοληθούμε λεπτομερώς με κάθε θέμα, με, κάτι, με κάθε άρθρο του κανονισμού για τη Μεσόγειο, χρειαζόμαστε ορισμένες ημέρες για να προσανατολιστούμε και να ετοιμαστούμε για τη συζήτηση. Ευχαρίστως να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Ευχαρίστως να εξετάσουμε λεπτομερώς όλα τα θέματα με τα εμπλεκόμενα μέρη. Και είμαστε στη διάθεσή σας για να αξιολογήσουμε την εφαρμογή του κανονισμού. Τέλος, όσον αφορά τις, επίσημε τις επιστημονικές ε, γνωμοδοτήσεις πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται τακτικά δηλαδή ε, στις αναλύσεις που κάνει για τα κράτη-μέλη πρέπει ε, από το 2002 αλλά και προηγουμένως να συμβουλεύεται τις επιστημονικές επιτροπές, πράγμα το οποίο πράττει ε, επιμελώς και σε ορισμένες περιπτώσεις αποφύγαμε να στείλουμε στις επιστημονικές ε, επιτροπές κείμενα όπου δεν θεωρούσαμε ότι γίνονται σεβαστά τα κατώτατα κριτήρια. Θέλαμε λοιπόν να μην αντιμετωπίσουν οι επιστημονικές επιτροπές καταστάσεις που ήταν δύσκολο να διαχειριστούν. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των ε, εγγράφων και ε, των ε, στοιχείων τα οποία διανύμουμε. Πρέπει να σας πω ότι οι απαντήσεις που δίνω σήμερα δεν είναι απαντήσεις οι οποίες ίσως είναι ικανοποιητικές για τους εκπροσώπους του κλάδου ή τους ευρωβουλευτές, αλλά αλλά εάν πρέπει να υπησέλθω σε λεπτομέρειες θα χρειαστεί να περάσουμε ώρες. Και όπως σας είπα είμαι έτοιμος να το πράξω και σήμερα η Επίτροπος μας είπε ότι είναι διαθέσιμη για να δώσει πληροφορίες πιο λεπτομερείς ε, σχετικά με την κατάσταση Μεσόγειο διότι αξίζει να ασχοληθούμε με συγκεκριμένη μορφή, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να αξιολογήσουμε την εφαρμογή του κανονισμού. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε. κύριε Λόβιν. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ επίσης και την προθυμία που δείξατε να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις εξαιρέσεις. Θα κάνουμε προφανώς την εργασία που πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια της Επιτροπής, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε και μια ανταλλαγή απόψεων, να λάβουμε άμεσα κάποιες πληροφορίες δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό άλλωστε θέλουμε για να κάνουμε και εμείς εδώ τη δουλειά μας. Έχω να κάνω ακόμη μία ερώτηση. Όταν έχουμε εδώ εκπροσώπους του κλάδου, θα ήθελα να απευθύνω σε αυτούς τους δύο κυρίους απευθεία την ερώτησή μου. Επί ποιες βάσεως λέτε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να βασίσει την απόφασή της. Πώς το λέτε αυτό, θα ήθελα να διευκρινιστεί αυτό, διότι τέτοιες καταστάσεις παρουσιάζονται συχνά και δεν πρέπει να φύγουμε με μία πικρή γεύση από αυτή τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην ίδια Τεχνική, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα στοιχεία για τη Μεσόγειο δεν είναι πλήρη για το 50 περίπου της 100 των αποθεμάτων που λαμβάνονται υπόψη. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο πέρσι στο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λένε ότι περίπου το 22% είναι ε, ε, από τα οποία υπερεκμεταλλεύονται ε, ένα 12% είναι καλά και το 50% είναι ε, στοιχεία τα οποία δεν είναι επαρκή. Αυτά ήταν η επίσημη παρουσίαση επιστημονικών στοιχείων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι. Επομένως, οι γνώσεις που έχουμε για τη Μεσόγειο είναι ελλειπείς, ανεπαρκείς, για τη διατήρηση και την κατάσταση κάποιων ε, αποθεμάτων. Ε, ισχύει η ασχή της πρόληψης. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω, ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφή στην αρχική μου παρέμβαση. Εμείς δεν ζητήσαμε ως περιφερειακή οργάνωση της Μεσογείου ε, παρατάσεις και εξαιρέσεις. Ζητούμε απλώς αξιολόγηση των επιπτάσεων του κανονισμού και σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, διότι ο κανονισμός αυτό σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο δεν αξιολογήθηκε ποτέ, ούτε εκ των προτέρων, ούτε το κάνει κάποιος αυτή τη στιγμή. Αυτό μόνον ζητούμε, να αξιολογηθεί ο κανονισμός για να μπορέσουμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο τροποποίησεων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ανδρέας Παρέα. Ε, δεν θα πω πολλά κύριε Πρόεδρε, ήθελα να κάνω μια πρόταση. Μια πρόταση επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι είναι διατεθειμένη ε, να μας δώσει όλες τις ε, ε δυνατές πληροφορίες και ο πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπε ότι η Επίτροπος, η κυρία Δαμανάκη, επειδή ο κλάδος ζητά αξιολόγηση επιπτώσεων, ε, και νομίζω ότι μετά από τρία χρόνια μπορούμε να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση και όπως έλεγα και εγώ πριν δεν ε, είπε κανείς ότι δεν θέλει κανονισμό ούτε είπε κανείς ότι δεν θέλουμε να ρυθμίζουμε πράγματα απλώς θέλουμε τη σωστή του εφαρμογή. Θα ήθελα να έρθει η κυρία Δαμανάκη να μας δώσει εξηγήσει και να δεσμευτεί να κάνει μια αξιολόγηση επιπτώσεων εάν μπορεί να το κάνει αυτό φυσικά. Η κυρία Ρόντους. Λοιπόν, το πρόβλημά μου δεν έχει λυθεί ακόμη διότι οι κυβερνήσεις, ε, μάλλον το Συμβούλιο, έχει συνενέσει και άρα οι κυβερνήσεις έχουν αναλάβει την υποχρέωση να διαθέσουν τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Όταν, ε, ε, αν άκουσα καλά τους εκπροσώπους του κλάδου, μας λέγουν ότι δεν τα κατάφεραν οι υπεύθυνε κυβερνήσεις, διαφορετικά δεν θα φτάναμε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτή την Επιτροπή ε, ε, να πρέπει να διορθώνουμε ε, τις παραλήψεις των κυβερνήσεων ιδίω όταν λάβει κανείς υπόψη πώς μας αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις και το Συμβούλιο και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά. Ο κύριος Σάντσες Περσέδο. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω κι εγώ. Εγώ θεωρώ ότι ο κανονισμός είναι απαραίτητος και αυτό που είναι σημαντικό είναι όταν ε, έχω θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη αλληλευτική πολιτική, να είναι και αποτελεσματική. Θα ήθελα να θέσω όμως δύο θέματα. Πρώτον, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η αλληλευτική μας πολιτική στην ίδια θάλασσα και με τους ίδιους πόρους, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, ώστε οι αρχές αυτές να τηρούνται και σε αυτές τις χώρες. Διότι αν δεν ισχύει αυτό, ε, ουσιαστικά θα δημιουργείται διαφορετική πολιτική στην ίδια θάλασσα με ίδιους πόρους για τα θέματα της εμπορικής πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε το πλαίσιο της ε, συνεργασίας με τις χώρες της Μεσογείου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα πράγματα και να έχουμε ε, καλή εφαρμογή του κανονισμού όχι μόνο σε άμεση επίπεδο αλλά και εν γέννη στην αλληλευτική πολιτική. Δεύτερον, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία είναι διαφορετικά. Το ένα αφορά την προσαρμογή στον κανονισμό. Ε, και ίσως δεν κατάφεραν όλοι να προσαρμοστούν, που σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι περίπλοκο και ίσως θα έπρεπε να το προχωρήσουμε εδώ το θέμα. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω καμία καθυστέρηση εδώ, αλλά από την άλλη υπάρχει και το γεγονό ότι ναι, μεν υπάρχει μια περίοδο τριών ετών, αλλά το ότι λήγουν οι εξαιρέσει στα τρία χρόνια δεν σημαίνει ότι δεν θα διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιε αντικειμενικέ δυσκολίε, ε, οι οποίε να μην οφείλονται απλώ ε, στο γεγονό ότι εξέπνευσε αυτή η προθεσμία των τριών ετών. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να τι λύσουμε. Εάν είναι πρόβλημα το μέγεθο των δικτυών και δημιουργούν προβλήματα και μειώνεται η αξία ενό είδου, τότε αυτό είναι ένα υπακτό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Από εκεί και πέρα, το μέγεθος των ε, δικτυών. Και εάν δημιουργεί προβλήματα και δεν μπορεί να γίνει αλλιεύση όπως προβλέπεται, και πάλι είναι ε, αντικειμενικό πρόβλημα σχεδιασμού και θα πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ε, θα πρέπει να δούμε δηλαδή κατά πόσο είναι αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε ανάγκη να το εξετάσουμε, διότι υπήρχαν οι εξαιρέσεις. Τα προβλήματα τα οποία αποτίθεται λοιπόν θα πρέπει να επιλύονται και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε και αποτελεσματικούς κανονισμούς. Πρόεδρος, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει πληροφορίε. Εγώ πραγματικά ενδιαφέρομαι προσωπικώ για το θέμα, διότι ασχολήθηκα με το θέμα αυτό, το ε, παρακολουθώ και θα ήθελα να συνεχίσω να το παρακολουθώ. Όχι για να επικρίνω τον ιονδήποτε, αλλά γιατί θα ήθελα να δω πώ εξελίσσεται η κατάσταση. Και αν μπορεί είτε με, μέσω μια σύνοψη ή μέσω μια πλήρους έκθεσης μπορεί να μας δώσει κάποιες πληροφορίες, ε, νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν όλους μας. Ε, Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει ένα νέο διάλογο με τον κλάδο, με το ράκ της Μεσογείου φαντάζομαι, και να συνεχίσει τις συζητήσεις και με τα κράτη-μέλη. Και επίσης υπάρχει αυτό που είπε ο κύριος Σάνσες Περσέδες, το οποίο το είπαν και άλλοι νομίζω, ότι θα πρέπει ε, και στις περιφερειακές οργανώσεις αλληλεία και στο ΚΑΤ και στην ε, περιφερειακή οργάνωση αλληλεία τη Μεσογείου θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα ώστε να προσπαθήσουμε να έχουμε συστάσεις οι οποίες ε, θα εφαρμόζονται. Ορισμένες αυτές έχουν εφαρμοστεί. Ε, το αν τις τηρούν τρίτες χώρες ε, ή μη είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά νομίζω ότι ο κανονισμός αυτή τη στιγμή είναι σωστός και προσπαθούμε τα ίδια μέτρα που εγκρίνονται εδώ σε εμά να εφαρμόζονται και αλλού. Το κατά πόσον γίνονται δεκτά ή όχι δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. έχουμε την υποχρέωση άλλωστε να είμαστε και το πρότυπο και είμαστε, να είμαστε οι πρώτοι που εφαρμόζουμε συγκεκριμένα μέτρα. Επομένως, ε, δεν θα το ε, θα συνεχίσουμε μάλιστα να είμαστε αυτοί που θα το κάνουμε πριν από όλες τις υπόλοιπε χώρες και από εκεί και πέρα να δίνουμε το σωστό παράδειγμα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εκεί και πέρα ε, να θέσουμε και το πλαίσιο της συζήτησης ε, με τους εκπροσώπους του κλάδου. τώρα το γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη παρουσίασαν προγράμματα διαχείρισης καθυστερημένα ή κάποια δεν παρουσίασαν τίποτε, αυτό μας το επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σημειώνουμε κι εμείς. Ολοκληρώνεται λοιπόν και αυτό το σημείο. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του δύο εκπροσώπου τη Περιφερειακή Οργάνωση Αλία για την παρουσία του εδώ. Και επειδή δεν υπάρχει κάτι ακόμα να συζητήσουμε εδώ σήμερα, ε, κλείνουμε τη συνεδρίαση μέχρι αύριο το πρωί. Θα ήθελα να σα ζητήσω να είστε στην ώρα σα, γιατί αύριο θα έρθει ο Προεδρεύον του Συμβουλίου και δεν θα ήθελα να είμαι εδώ μόνη μαζί του. Θα ήθελα να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερου ε, βουλευτέ παρόντε ε, για να προσπαθήσουμε να ε, υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει